la sovrapposizione di un Sanremo, tutto il PPS era a Palermo. Okay, good morning, ladies and gentlemen. Can we make a start? We're running a few minutes late. Μπορούμε να ξεκινήσουμε καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Επαναλαμβάνω, ορίσατε στην Επιτροπή Αλίας. Ε, μου ζητήθηκε να αντικαταστήσω την ε, Κάρμεν Φράγκα σήμερα η οποία δυστυχώς έχει ε, κάποια προβλήματα υγείας ε, που αφορούν μέλη της οικογένειάς της. Ε, θα μπορέσει να είναι μαζί μας από την Τετάρτη και μετά. Οπότε έχουμε τρεις ε, σημαντικές αλλαγές στη σημερινή ημερήσια διάταξη Οι τέσσερις ενδεχομένω αλλαγές. Είναι που, κάτι που περιπλέκει τα πράγματα. Καταρχήν, ένα αίτημα της ε, ε, Κάρμεν Φράγκα της Προέδρου για ψηφοφορία του νέου πρωτοκόλου με τη Μικρονησία. Αυτό θα πρέπει να αναβληθεί μας ζητάει ε, και τονίζει όχι γιατί είναι πόνο εισηγητής, γιατί έχουμε και μια άλλη εισήγηση σήμερα το πρωί την οποία θα εξετάσουμε ε, με τον ίδιο εισηγητή, αλλά γιατί η ίδια η Μικρονησία αποφάσισε να μην επικυρώσει το πρωτόκολλο παραμετά τις εκλογές, οι οποίες θα γίνουν στο τέλος του Μαΐου. Οπότε η κυρία Φράγα θεωρεί ότι δεν είναι κατάλληλο να ψηφίσουμε το ε, του πρωτοκόλου μετά από την Μικρονησία, από την, ε, δεν μπορούμε πριν να επικυρώσει η Μικρονησία, δηλαδή να ψηφίσουμε εμείς. Ύστερα, ο κύριος Άντεκ ο οποίος ε, ε, είναι απαραίτητο να είναι σε μια άλλη συνεδρίαση στις 10.30. Στο σημείο 8 έχουμε ένα νέο πρωτόκολλο για τον καθορισμό της χρηματικής αντιπαροχής μεταξύ Σεϊχελών και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε πρέπει να το δούμε αυτό τώρα, μετά από το 5 και το 6. Και ύστερα ζήτησε ο κύριος Χάγκλεν να, να σας πω ότι δεν μπορεί να είναι παρόν στη συνεδρίαση για τη συμφωνία με το Μαρόκο σήμερα ε, και συνεπώς με, μια, με την επέκταση του σχετικού πρωτοκόλου ζητήθηκε λοιπόν να αναβληθεί και αυτό το θέμα. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι ε, θα είχε συζητηθεί στην αυριανή συνεδρίαση, αλλά τώρα ακυρώθηκε πλήρως. Οπωσδήποτε αύριο ταξιδεύετε προς τις Ασόρες κανονικά, που σημαίνει ότι θα φεύγατε στις 10 το πρωί από τη συνεδρίαση, ενώ τώρα ακυρώνεται πλήρως η αυριανή συνεδρίαση. Και ε, δεν έχουμε χρόνο να συζητήσουμε την συμφωνία με το Μαρόκο θα ήθελα να πληροφορήσετε όλους τους απόντες συναδέλφους σήμερα ότι αύριο το πρωί δεν έχουμε συνεδρίαση. Λοιπόν, με αυτές τις προσαρμογές σας προτείνω να καταρτήσουμε την ημερήσια διάταξη έτσι όπως την προτείναμε. Η... Θα υπάρχει web stream στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αυτή της σημερινή μα συνεδρίαση. Υπάρχει μια ε, δυνατότητα παρακολούθησης της ε, Επιτροπής Λίμπερ. ζήτησε λοιπόν στην απουσία της αν είναι δυνατόν να ε, δούμε το δικό της σημείο στην ημερήσια διάταξη, το οποίο περνάει κανονικά πριν από τις 10, να το καθυστερήσουμε. Έχουμε την έκθεση του κυρίου Καπούλα Σάντες, παραδείγματος χάρη, που μπορούμε να το δούμε πριν η κυρία Γιώτοβα Φαντάζομαι ότι θα είναι εδώ πριν να ε, δούμε το σημείο στην ημερήσια διάταξή της, δηλαδή δεν χρειάζεται νομίζω να κάνουμε άλλη αλλαγή στην ημερήσια διάταξη. Ωραία. Λοιπόν, μετά από αυτή την αναδιάρθρωση της ημερήσιας διάταξης, ας περάσουμε στο σημείο 2 που είναι η έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων της 15ης και 16ης Μαρτίου 2011. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις και δεν έχουμε ακούσει αντιρρήσεις πριν από την Επιτροπή, θεωρούν συγκεκριμένα. Για τις ανακοινώσεις του Πρόεδρου, θα ήθελα να υπενθυμίσω στα μέλη που φεύγουν αύριο για την αντιπροσωπεία η οποία πηγαίνει στην Πορτογαλία και στις Ασόρες ότι το ε, σημείο που συναντιόμαστε αύριο το πρωί είναι 9 και 4 αύριο το πρωί στο, εκεί που είναι η Σοφέρ 10 ε, και 4 λοιπόν γιατί η αναχώρηση είναι στις 10 και μισή η αναχώρηση του λεωφορείου στη συνέχεια έχουμε το σημείο το οποίο αναβλήθηκε δηλαδή την ψηφοφορία με τις για τις ομόσπονδες πολιτείες της Μικρονησίας. Περνάμε στις άλλες ψηφοφορίες λοιπόν, η οποία είναι στο σχέδιο έκθεσης ε, ε, για τα μέτρα που λαμβάνει το κράτος λιμένα για την πρόληψη, αποτροπή και εξάλληψη της παράνομης λαθρέας και άναρχης αλίας. Ε, είχε προταθεί η έκθεση της κυρίας Φράγκα στο, ε, στο Συμβούλιο για απόφαση του Συμβουλίου στην, ε, στο άρθρο, σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 6α ε, παραπέμπεται εκεί, ζητείται η γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου και ζήτησε έγκριση από το Κοινοβουλίο με, μια, με ένα σχέδιο έκθεσης, το οποίο ε, ε, την έκθεση αυτή προετοίμασε ο ε, δικηγόρος της νομική ε, νομικής υπηρεσίας. Η κυρία Φράγκα στις 15 Μαρτίου παρουσίασε μια άλλη, ένα άλλο σχέδιο έκθεσης. μόνο μία τροπολογία κατατέθηκε και ήθελα να υπενθυμίσω στην Επιτροπή ότι αυτή η έκθεση ε, ε, προτείνεται βάσει του άρθρου 2, 6α της συνθήκης όπου το Κοινοβούλιο μπορεί να δώσει ή να μην δώσει τη σύμφωνη γνώμη του. Ε, και πρέπει να πούμε ότι υπάρχει ε, ενώ κανονικά δεν δεχόμαστε τροπολογίε σε μια πολύ περιορισμένη βάση αν υπάρξουν τροπολογίε επί τη διαδικασία και όχι επί τη ουσία, είναι δυνατόν να κατατεθούν ε, έτσι κατατέθηκε η τροπολογία του κυρίου Ασένα. Επίση, υπενθυμίζω ότι τα μέλη που έχουν αντίθετη σχέση, ε, θέση με την θέση του εισηγητή μπορούν να καταψηφίσουν το σχέδιο ψηφίσματο. μετά από αυτές τις ανακοινώσεις μπορούμε να περάσουμε στην ψηφοφορία ε, υπάρχει μια τροπολογία του κύριου Ασένας και μια πρόταση προφορικής τροπολογίας από τον εισηγητή και ο κύριος Κάδικ θα μας, πει, την, θα μας ε, διαβάσει την προφορική τροπολογία. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στην τροπολογία που κατατέθηκε θα ήθελα να υπάρξει μια προσθήκη. Γράφεται στην καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προωθήσει ενεργά την υπογραφή, επικύρωση και εφαρμογή της συμφωνίας σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνει το κράτος λιμένα για την πρόληψη, αποτροπή και εξάλληψη της παράνομης λαθρέας και άναρχης αλίας στο πλαίσιο των εμπορικών συμφωνιών. Σε αυτό το σημείο να προσθεθεί των περιφερειακών οργανώσεων διαχείρισης της αλληλείας και μετά συνεχίζουμε των συμφωνιών αλληλευτικής σύμπραξης και της αναπτυξιακής πολιτικής της Ένωσης. Αυτή είναι, αυτό είναι η προφορική τροπολογία την οποία θα ήθελα να προσθέσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κάδεκ, υπάρχει κανείς που έχει αντίρρηση σε αυτήν την προφορική τροπολογία. Εφόσον όχι, έχετε τις κάρτες σας για να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Κύριε Σάντες. And then we will move to the votes. Okay. Ωραία λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Ομοφωνία. και επί της νομοθετικής προτάσεως ψηφίζουμε τώρα ο σύνολο, άρχεται η ψηφοφορία, ψήφισαν όλοι, πέρας. Και εδώ έχουμε ομοφωνία. Συγχαρητήρια λοιπόν στον, στην συγκητία. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα, ε, έχοντας υπόψη ε, τις, ε, το, τις αλλαγές που κάναμε στην ημερήσια διάταξη, μπορούμε να περάσουμε στο θέμα 8 που είναι η έκθεση του κυρίου Κάντεκ για το νέο πρωτόκολλο για τον καθορισμό των αλλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη Συμφωνία Αλλιευτικής Σύμπραξης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Δημοκρατίας των ε, Σεϊχελών. Στις 14 Ιανουαρίου ε, ε, πήρε, έλαβε το Κοινοβούλιο την αναπομπή από το Συμβούλιο και από την ε, ημερομηνία αυτή και μέχρι τις 26 Ιανουαρίου ε, ανατέθηκε η εξέταση αυτής της Επιτροπής στο σχέδιο έκθεσης. Το Μάρτιο έγιναν ε, οι εξετάσεις των αλλαγών του πρωτοκόλου και σήμερα ο εισηγητής προς, μας παρουσιάζει το πρωτόκολλό του και οπότε σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν σας ευχαριστώ που μου δώσατε τη δυνατότητα να πάω στην επόμενη επιτροπή βάζοντας ε, αυτό το σημείο νωρίτερα στην ημερήσια διάταξη. Δυστυχώς δεν είναι πολλοί παρόντες ε, βουλευτές που ε, ενδιαφέρονται για τη συμφωνία με τις Σεχέλες. Ήταν τρεις συμφωνίες μαζί με το Μαρόκο και την Μαυριτανία ε, θα ήθελα να σας παρουσιάσω γρήγορα αυτή την έκθεση που την βρίσκεται σε διάφορες γλωσσικές εκδοχές στο Κοινοβούλιο ε, τα ε, πλοία διέπονται από μια συμφωνία που ισχύει από, τον, από τις 18 Ιανουαρίου μέχρι τις 15 Μαρτίου και βλέπετε ότι έχουμε ξεπεράσει την ημερομηνία. Ήρθε δηλαδή η ώρα να το διεκπαιρεώσουμε αυτό το θέμα. Έγιναν διαπραγματεύσεις μεταξύ της Δημοκρατίας των Χελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπογράφηκε ένα πρωτόκολλο για τρία χρόνια που θα αρχίσει με έναρξη ισχύω στις 3 Ιουνίου. Ε, οι Σεχέλες ε, έχουν μια περιοχή 14.000 τετραγωνικών μέτρων ε, και αφορά τον τουρισμό και την αλία οι 15% ε, του ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος είναι αυτή η δραστηριότητα, 17% του ενεργού πληθυσμού συνολικά ασχολείται. Η αλία λοιπόν και η μεταποίηση των νυχθείων είναι πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία για την οικονομική δραστηριότητα του αρχιπελάγους. 400 είναι οι ενότητες, και ε, υπάρχουν ε, πλοία τα οποία, ε, αυτά τα 400 πλοία αλλιεύουν σε αυτή την περιοχή. Η συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση αφορά έναν στόλο επίσης ασιατικό ο οποίος έχει πλοία με σημαία της, των Σεχελών και είναι μια joint venture. Έχουμε επίσης ένα σημαντικό όγκο αλίας, πάρα πολύ σημαντικό για την αγορά μας. Το νέο πρωτόκολλο προβλέπει 7,8 εκατομμύρια ευρώ ε, για, για τρία χρόνια για το σύνολο των αλλιευτικών δραστηριοτήτων και έχουμε ένα ποσό 3,38 εκατομμυρίων ε, ευρώ και 2,22 εκατομμύρια ευρώ υποστήριξη από πλευρά Σέχελων για, σαν επιπρόσθετο ποσό ε, για την άσκηση της ε, ε, θαλάσσιας για την άσκηση της αλίας στην ίδια ζώνη. Πρέπει να πούμε επίσης ότι ο Ευρωπαϊκός Στόλος έχει διάφορες δυνατότητες με 48 πλοία τα οποία από το 2007 έχουν εγκαταλείψει αυτή την πολύ επικίνδυνη ζώνη, όπως γνωρίζετε είναι επικίνδυνη λόγω της πειρατείας. Και οπότε τα αλλιεύματα είναι πολύ χαμηλότερα από 300.000 τόνους το χρόνο. Ε, υπάρχουν γρηγροί και παραγάδια. Ε, πρέπει να γίνεται μια επιθεώρηση ε, πάρα πολύ έντονη και γι' αυτό υπάρχει, ζητήθηκε μία έκθεση ε, για την πειρατεία στην περιοχή. Ε, ανάμεσα στο 2006 και το 2009 υπήρχαν αρνητικές επιπτώσεις στην αλία και στην συνεργασία μεταξύ ΕΕ και Σεχελών. Υπάρχει η επιχείρηση Αταλάντη που θα γνωρίζετε που αφορά την καταπολέμηση της πειρατείας το ιδεώδες βεβαίως θα ήταν να ξαναφτάσουμε στην προηγούμενη κατάσταση, ούτω ώστε να μπορούν όλοι να λιεύουν σε αυτή την αποκλειστική ζώνη. Σε ό,τι αφορά τα αποθέματα τα αλλιευτικά, η αλληλεία έχει τρία είδη ψαριών, τον αλμπακόρ, το λιστάο και το πατόντο. Αυτά αφορούν το λιστάο ειδικά, ε, είναι ένα είδος ε, που ε, καλύπτει ένα 50% των τιμών της πώλησή του και ε, έχουμε ένα πολύ μικρό ποσοστό των αλμπακόρ που είναι 1% περίπου, οπότε είναι εντελώ περιθωριακό. Τα τελευταία ε, χρόνια βλέπουμε ότι υπάρχει πλήρης εκμετάλλευση του πατόντο, του ξηφία ε, και του αλμπακόρ σε μια πολύ μικρότερη κλίμακα το θέμα αυτό μας ανησυχεί γιατί συμμεριζόμαστε με τις αρχές αυτήν την ανησυχία. Υπάρχει αλίευση γόνου, ε, κάτι που μας ανησυχεί εδώ και πολύ καιρό, καθώς και τον οργανισμό ο οποίος επαγρυπνεί να μην ε, γίνεται υπεραλίευση του γόνου. Γνωρίζουμε λοιπόν ότι ε, υπάρχει αυτή η κακή πρακτική υπάρχουν αποφάσεις οι οποίες έχουν ληφθεί για να γίνεται η αλία μόνο από δηλωμένα γρηγρή και παραγάδια ε, που έχουν επίσημες άδειε αλίας ούτω ώστε να μην ε, αλλάζουν τα ποσοστά των αλιευμάτων. Ε, σας υπενθυμίζω ότι υπάρχουν αλίες οι οποίοι έχουν ε, γειτονικές, αλιεύουν σε γειτονικές ζώνες με παρόμοια ε, σκάφη και έχουμε 230 άδειες για τους ε, αλείς των Σεχελών, 760 άδειες για την Ευρώπη. Και βλέπετε ότι ε, μέσα στην εξέλιξη της αλίας υπάρχει μια ποσόστοση η οποία πηγαίνει προς την ίδια κατεύθυνση. Τα ευρωπαϊκά πλοία τα οποία έχουν άδεια να αλιεύουν στις Σεχέλες έχουν και παρατηρητές μαζί τους οι οποίοι υπάγονται στην φύση που ασκεί έλεγχο αποτελεσματικό και ο έλεγχος αυτός μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε μια παρουσία στον ειδικό ε, ωκεανό και να ε, κατοπτεύουμε. Επίσης έχουμε δύο ναυτικούς από τις Σεϊχέλες οι οποίοι μαζί με τον πλειοκτήτη είναι παρόντες στα πλοία και ε, οι Σεχέλες προτείνουν έναν κατάλογο όπου ε, ε, πλοίων όπου μπορούν να ε, πάνε οι παρατηρητές στα ύδατα των Σεχελών μέσα στα πλαίσια της συμφωνίας διαρκεί και γίνεται διαρκής αλληλεία υπάρχει μία ρήτρα διακοπής πώς προβλέπετε να εφαρμοστεί αυτή η ρήτρα διακοπής μόνο αν υπάρξει παραβίαση των δικαιωμάτων. Και αυτή η διακοπή επίσης είναι δυνατόν να γίνει αν δεν υπάρχει σεβασμός των συνθήκων εργασίας και των κανόνων εργασίας που θεσπίζουν οι αρμόδιες αρχές. Και εδώ περικλείται και η αλληλεία. Υπάρχουν πολλές πηγές ανησυχίας, οι οποίες όμως δεν θέτουν ένα αμφιβόλο την ίδια τη συμφωνία. Η πειρατεία, όπως σας είπα και πριν, ε, εμποδίζει την αλληλεία. Οι Σεϊχέλες είναι η μόνη κυβέρνηση, υπογραμμίζω, η οποία δέχεται να δικάσει τους πειρατέ και που θεωρεί θετική την καταπολέμηση της πειρατείας. Η εργασία αυτή γίνεται από κοινού με τις αρμόδιες αρχές οι οποίες δικάζουν τους πειρατές και οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να τους καταδικάσουν. Ε, ένα 70% της αλίας του τόνου γίνεται από τα γρηγρή και ε, πρέπει να επαγρυπνούμε για την γιατί υπάρχουν ε, πάρα πολλές ε, εκδηλώσεις ε, υπεραλίευσης του γόνου. Γι' αυτό πρέπει να ελέγχουμε πάρα πολύ καλά την περιοχή και το πράττουμε. Το 2010, 69% των αλλιευμάτων των Σεχελών γινόντουσαν από τα ευρωπαϊκά σκάφη. Και άλλες χώρες είναι η Ιαπωνία, η Κίνα που αλλιεύουν επίσης. Και επαναλαμβάνω κάθε φορά την ανησυχία μου την οποία γνωρίζετε ορισμένοι όπως η ε, Κινέζοι αλληλείς παραδείγματος χάρη υπεραλλιεύουν. Ε, χωρίς άδεια ψαρεύουν μεγάλες ποσότητες και πρέπει λοιπόν να είμαστε παρόντες, να υπάρχουν πάντα ευρωπαϊκά πλοία στην περιοχή για να ε, διατηρείται η ισορροπία και ο έλεγχος του όλου συστήματος. Η συμφωνία αυτή είναι αποτελεσματική διότι επιτρέπει την δυνατότητα ανάπτυξης του ευρωπαϊκού στόλου και δίνει θέσεις εργασίας και στις αιχέλες οι οποίες συμβαλούν στην ανάπτυξη ε, της χώρας αυτής μπορούν να αναπτύξουν μια υπεύθυνη αλληλεία. Ε, η προηγούμενη, ο προηγούμενος τύπος δεν, ε, αλληλείας δεν προστάτευε ικανά το γόνο και τα αλλιεύματα. Σήμερα με αυτή τη συμφωνία υπάρχει συμμετοχή της ευρωπαϊκής αγοράς, κατασκευή της κονσέρβας του τόνου και στις Εχέλες υπάρχει μια έντονη δράση, δραστηριότητα γύρω από αυτόν τον τομέα Νομίζω ότι και οι δύο πλευρέ έχουν μεγάλο όφελο, και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Σεχέρε από αυτή τη συμφωνία. Θα ήθελα να είναι πλήρω πληροφορημένο το Κοινοβούλιο για, τις, για τα συμπεράσματα τη Μικτή Επιτροπή και μέλη του Κοινοβουλίου να μπορούν να παραβρεθούν σε αυτέ τι συνεδριάσει. Το ζήτησα ήδη και ζήτησα και μία, ένα σχέδιο έκθεση για το 2014 για την εφαρμογή αυτού του πρωτοκόλου, ώστε να μπορέσουμε να προετοιμάσουμε στη συνέχεια το επόμενο πρωτόκολλο. Η Επιτροπή Προπολογισμού και ε, σε σχέση με τα σημεία τα οποία έθεσε η ε, υπέβαλε Επιτροπή Ανάπτυξης η οποία αποφασίζει για τα σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν με προϋπολογισμό από την ε, κοινότητα ειδικά για την Βικτόρια νομίζω ότι θα πρέπει να επιληφθούμε αυτού του σχεδίου και πιστεύουμε ότι τα ποσά τα οποία καταβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δαπανούνται υπέρ των αλλιέων, υπέρ των αλλιευτικών δραστηριοτήτων. Αυτό πρέπει να το, το έχουμε ελέγξει αρκετά ε, ενδελεχώς και βλέπουμε ότι ε, δαπανούνται ε, τα ποσά για την άσκηση της αλίας στις κατάλληλες ζώνες. Η SFA είναι πάρα πολύ ικανή και αποτελεσματική, κάτι το οποίο δεν ισχύει σε όλες τις περιοχές του Ειρηνικού και του Ατλαντικού. Ζητήσαμε ένα πρωτόκολλο, είπαμε, καινούργιο από 2014 και αυτό είναι σε απάντηση ε, ε για τα, στα αιτήματα των δύο επιτροπών. Ε, Επίσης υπάρχει μια γνωμοδότηση την οποία θα υποβάλουμε ως Κοινοβουλευτική Επιτροπή αυτό είναι γενικά το περιεχόμενο της έκθεσής μου αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, σας καλώ να υποβάλλετε σχόλια ε, και υπάρχουν ε, ενδείξεις, έχουμε ακούσει ότι είναι πάρα πολύ ικανοποιημένε οι αρχές της δημοκρατίας των Σεχελών από τις προτάσεις που υποβάλαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Καντέκ για αυτή την ε, Καλή παρουσίαση. Πρώτα απ' όλα η κυρία Ανδρέας ζητάει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ως σκιώδης εισηγήτρια απλώς θα ήθελα να πω ότι αυτά τα οποία είπε ο κύριος Καντέκα αντικατοπτρίζουν την, κανονική, την ισχύ κατάσταση. Νομίζω ότι ήταν υποφελής και γιατί δύο μέρη συμφωνία αυτή. Είναι η πιο σημαντική μετά από αυτό με τη Μαυριτανία η πιο παλιά και είναι πάρα πολύ χρήσιμη και για τον ευρωπαϊκό αλευτικό στόλο και διότι ε, έχει πολλά ωφέλη για όλους. Από την πλευρά της αλίας πρέπει να πω ότι είναι μία συμφωνία πλαίσιο δεδομένου ότι πληρεί τα κριτήρια αηφορίας, δέχεται την επιστημονική συνεργασία, τους παρατηρητές και εισαγάγει και το θέμα του να αλλιεύουν στα σκάφη και τοπικοί αλλιείς. Η χώρα επωφελείται από αυτή τη συμφωνία που μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για την περιοχή και συμπεριλαμβάνει και ένα σημαντικό στοιχείο που είναι η ρήτρα τήρησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων με δικαίωμα αναστολής των δραστηριοτήτων εάν δεν τήρονται. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο ενισχύει τις προσπάθειες εκδημοκρατισμού της περιοχής και αν οι εργαζόμενοι αποτελέσουν αντικείμενο εκμετάλλευσης μπορούν να προσφύγουν στο Διεθνές Γραφείο Εργασίας. Απ' την άλλη ε, υπάρχει και η έννοια της πειρατείας που είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι, μιλάμε για περιοχή επικίνδυνη. Οι πειρατές δημιουργούν προβλήματα και για τους ολιευτικούς μας αλλά γενικότερα από την ε, αλληλεία είναι και θέμα ασφάλειας με τις ε, επιχειρήσεις τύπου Αταλάντη, νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε μια πολύ καλή συμφωνία για την περιοχή, για την καταπολέμηση της ε, ε, πειρατείας που είναι πάρα πολύ σημαντική για την ασφάλεια της περιοχής. Πιστεύω λοιπόν ότι πρόκειται για κάτι το πολύ σημαντικό για την περιοχή, για όλη τη ζώνη, για τη χώρα, για την αλληλεία, για την ασφάλεια. Επίσης, για μας είναι θέμα ισορροπίας της αγοράς και όπως είπε και ο κύριος Καντέκ, αποτρέπει την παρουσία τρίτων χωρών που δεν σέβονται τους κανόνες, μεταξύ άλλων τους κανόνες αηφορίας όπως και εμείς. Ευχαριστώ. Θα υποστηρίξουμε την έκθεση λοιπόν αυτή. Σας ευχαριστώ κυρία Ζαντρές. Κυρία Λοβέ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Καντέ και την έκθεση. Έχω τέσσερις πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις που με απασχολούν. Δεν διάβασα την ίδια την έκθεσή σας. Διερωτώ με, δεδομένου ότι υπάρχουν λιγότερες αλλιευτικές δυνατότητες εξαιτία της πειρατείας τα τελευταία χρόνια, σημαντικά λιγότερες, και εδώ βλέπω ότι έχουμε στο ε, νέο πρωτόκολλο 48 νέα αλλιευτικά σκάφη τράτες και 12 με παραγάδια, διερωτώ γιατί έχουμε συμπληρωματικά αλλιευτικά σκάφη στο νέο πρωτόκολλο, δίδοντας περισσότερες ε, άδειε ενώ έχει μειωθεί η αλλιευτική δραστηριότητα. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν περί τίνος πρόκειται. Αν μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει, η συμφωνία αυτή προβλέπει και κάτι προσωρινές συμφωνίες εάν δημιουργήσουν μεγάλη απειλή οι δραστηριότητες των πειρατών. Ίσως θα μπορούσε η Κομισιόν να μας εξηγήσει περί τίνος πρόκειται. Τρίτη ερώτηση. Γίνεται με τα παραλιεύματα. Σύμφωνα με την έκθεση του κυρίου Καντέκ. Ο... Ένα από τα απειλούμενα είδη είναι ο μεγαλόθελμος τόνος. Θα ήθελα να μου πει τι γίνεται με τις δραστηριότητες παραλίευματο. I see that and I understand. Από ό,τι καταλαβαίνω υπάρχουν πολλές δυνατότητες δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης και στην ε, μεταποιητική βιομηχανία και όλες στις Σεϊχέλες. Ό,τι γίνεται έχει επίσης ως στόχο την προώθηση δραστηριοτήτων στον τομέα αυτό. Ποιες είναι οι εξελίξεις, τι γίνεται με τον τομέα της λίας, τον τοπικό στις Σεϊχέλες, αναπτύσσεται ή μόνο τομέα της κονσερβοποίησης και της μεταποίησης επωφελείται από τη συμφωνία αυτή. Αυτές είναι οι ερωτήσεις μου. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Λόβα. Θα ήθελα κι εγώ όσον αφορά την πειρατεία να πω το εξής. Έχουν συλλάβει αλλιευτικά σκάφη κοινοτικά οι πειρατές, θα μπορούσε να μας το πει η Κομισιό. Ε, κρατή, ε, συνελήφθησαν κάποια, πληρώθηκαν λίτρα, ποιος τα πλήρωσε, έχετε πληροφορίες. Τώρα, από την Κομισιό ο κύριος Αλεξάνδρου από την ΜΑΡΕ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πριν απαντήσω στις διάφορες ερωτήσεις που κάνουν οι διάφοροι συναδελφοί σας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Καντέκ, για αυτή την εξαιρετική έκθεση, διότι πολύ σύντομα ανέφερε τα θεμελιώδη στοιχεία περιέχοντες από το πρωτόκολλο και χωρίς να μπει σε λεπτομέρειες, πρέπει να πούμε ότι ποιοτικά πρόκειται για μία μεγάλη πρόοδο σε σχέση με τα προηγούμενα πρωτόκολλα. Κύριε Καντέκ, επιμείνατε για τα κύρια θετικά σημεία αυτής της ε, νέας συμφωνίας και τα συμμεριζόμαστε και εμείς μαζί σας. Επίσης, υπογραμμίσατε ποια είναι η πρόκληση που τίθεται για την περιοχή, η πειρατεία πολύ μεγάλη πρόκληση, δεδομένου ότι πρόκειται για δραστηριότητα η οποία απειλεί την ασφάλεια των λιευτικών σκαφών που θέλουν να επιχειρούν στην περιοχή με νόμιμο τρόπο, όχι μόνο στην περιοχή των Σεϊχελών, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του Δυτικού Ινδικού ωκεανού. Αυτό το φαινόμενο θεωρούμε ότι είναι ένα πραγματικό ε, πλήγμα για την περιοχή και η Αταλάντη ξέρουμε ότι επέκτασε δραστηριότητες νοτίως για να μπορέσει να συμπεριλάβει και την εποπτεία των υδάτων της, ε, των Σεϊχελών. Υπάρχει ένα άλλο τρομερό πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να αναφέρω. Η ανάπτυξη άναρχης ε, αλίας. Όχι μόνο στην περιοχή των Σεϊχελών, αλλά και σε άλλες παράκτιες χώρες και παρά το γεγονός ότι κάποιοι δεν δίνουν μεγάλη σημασία σε τέτοιες συμφωνίες, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ελέγχουν πολύ σωστά τον λευτικό μας σκητό, δεδομένου ότι υπάρχουν πολλοί άλλες μικροί αλλιευτικοί στόλοι πι ε, λάμδα α που αλλιεύουν με καταστροφικό τρόπο και άναρχο. Πρόκειται λοιπόν για το δεύτερο πλήγμα το οποίο υφίστανται οι χώρες ε, του Δυτικού Ινδικού Ωκεανού. Ως υπεύθυνο λοιπόν της Επιτροπής για αυτά τα θέματα έπρεπε να σας αναφέρω αυτά τα δύο σοβαρά προβλήματα τα οποία ε, πλήττουν την ε, ε, περιοχή. Θα προσπαθήσω τώρα να δώσω κάποιες απαντήσεις σε ερωτήσεις τις οποίες έκανε και η κυρία Λέβιν ε, δίδοντάς σας αντικειμενικές απαντήσεις. Τις δυνατότητες αλίας ήμουν σίγουρος θα έθετε το θέμα αυτή κυρία Λέβη. Θα προσπαθήσω να είμαι πάρα πολύ ε, σαφής. Στις ε, συμφωνίες για τον τόνο, όπως ξέρετε, δίδονται άδειες ειδικέ και είπατε πάρα πολύ σωστά ότι έχουμε δώσει κάποιες άδειες ε, για τον τόνο. Από 40 ε, έγιναν 48 για τις στράτες του πρωτόκολλου. Υπάρχει λοιπόν αύξηση. Επίσης διαπιστώσατε ότι η χωρητικότητα αλίες που είναι δείκτης για το σύνολο της αυτοδικής δραστηριότητας, κυρίως για την ε, καταβολή τιμής για την πρόσβαση, μειώθηκε πάρα πολύ, διότι διαπιστώσαμε ότι εξαιτίας της πειρατείας τα αλλιεύματα είχαν πάρα πολύ μειωθεί το 2008 και 2009, ενώ έχουμε μια κάποια ανάκαμψη το 2010. Βάσει λοιπόν αυτών των εξελίσεων και για να μπορέσουμε να έχουμε μια υπεύθυνη διαχείριση των δημοσίων πόρων, δεδομένου ότι πρόκειται κυρίως για δημόσια χρήματα, τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων, για να κάνουμε λοιπόν σωστή, χρηστή διαχείριση αυτών των πόρων, συνεισφέραμε στην μείωση της χωρητικότητας ε, αναφοράς. Γι' αυτό βρίσκεται να υπάρχει αυτή η αντίθεση, δηλαδή αύξηση του αριθμού των αδειών από τη μια και από την άλλη μείωση της χωρητικότητας αναφοράς. Θα ήθελα εξάλλου να υπενθυμίσω ότι ο αριθμός που αναφέρεται εδώ είναι ο ανώτατος και σε πολλές περιπτώσεις ποτέ δεν φτάνει ε, σε αυτό τον αριθμό. Δηλαδή, αριθμός ετήσεων ε, αδειοδότησης και χορήγησης. Χρησιμοποιούνται λοιπόν ε, οι άδειε κατά το αριθμό, αλλά δεν χρησιμοποιούνται Τώρα, όσον αφορά αυτό το πρότατα temporis, δεν πρόκειται για ένα τέχνασμα για να πληρώνουν πολύ λιγότερα χρήματα όσον αφορά την προκαταβολή εφοπλιστές. Πρόκειται για ένα μηχανισμό ο οποίος προβλέπεται και χορηγείται με την σύμπραξη των αρχών της Αιχέλης, διότι δεδομένου ότι υπάρχει κάποιος προβλεπόμενος κίνδυνος, ενδεχομένως δηλαδή αύξηση της πειρατείας και σε αυτή την περίπτωση όχι μόνο στα ύδατα των Σεϊχελών δεν θα αλλιεύουν τα λεφτικά αλλά όλη την περιοχή. Δεδομένου λοιπόν ότι υπάρχει αυτός ο ενδυνάμει κίνδυνος και δεδομένου ότι αποχωρούν αυτά τα ε, σκάφη, καταβάλλεται αυτό το ποσό το προράτα τέμπορης, η προκαταβολή αυτή, και δεν πρόκειται για μία εξαίρεση, αλλά για να ληφθεί υπόψη αυτή η ιδιάζουσα κατάσταση στην οποία ενδεχομένως θα μπορούσαν να ευρεθούν κάποια σκάφη τα οποία αναπτύσσουν τις αλληλευτικές δραστηριότητε στον ε, Δυτικό Ινδικό ωκεανό. Και βεβαίως δεν πρόκειται για ανοιχτή πόρτα, διότι η αρμόδια αρχή για την αλία των Σεϊχελών είναι πάρα πολύ δυναμική, παρακολουθεί εκ του σύναγκη όλε τι δραστηριότητε, δεδομένου ότι υπάρχει παρακολούθηση 24 ώρε 24 ώρο με τα συστήματα VMS, τα σκάφη. Η αρχή λοιπόν παρακολουθεί εκ του σύναγκη, επαναλαμβάνω τι αλληλευτικέ δραστηριότητε και είναι σε θέση να δει στην οθόνη αν το αλληλευτικό σκάφο αποχωρεί οριστικά από την ε, αλληλευτική περιοχή των Σεϊχελών. Αν αποχωρήσει ε, το αλευτικό σκάφος και επανέλθει και πάλι θα κάνει, ε, πρέπει να υποβάλει αίτηση για νέα άδεια και θα πρέπει τότε να, καταβάλει, να καταβληθεί το σύνολο του ποσού που ε, προβλέπεται. Ξέρω ότι επίσης προσδίδει μεγάλη σημασία στην τοπική αλληλεία σε επίπεδο βιοτεχνίας εμείς τα λέγαμε. Στις 9 και 11 Φεβρουαρίου υπάρχει έγγραφο το οποίο εγώ επικύρωσα και στην σελίδα 3, στην παράγραφο 2-3, για τα θέματα της πολιετούς μήτρας που είναι η συμφωνία για την παρακολούθηση της υποστήριξης στον κλάδο αυτό θα δείτε για το 2011, 12 και 13 προβλέπονται πολύ σημαντικά ποσά για την βελτίωση, παραθέτω, της διαχείρισης της ε, τοπικής αλληλείας σε επίπεδο βιοτεχνίας και σε επίπεδο βιομηχανίας. Και θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια οι αρχές στις αιχέλες καταβάλουν προσπάθειες ώστε να μπορέσει να αναπτυχθεί και η, η δραστηριότητα των τοπικών αλλιέων Και εμείς βεβαίως δεν μπορούμε να είμαστε αντίθετοι. Για το 2011 έχουμε 319 εκατομμύρια, ε, συγγνώμη, 1788 και 1.599 για τα έτη 11, 13. Προβλέπετε λοιπόν με ακρίβεια το ποσό το οποίο θα δοθεί στην βιομηχανία την, ε, την βιομηχανική αλία και στην αλία την τοπική. Σημεριζόμαστε λοιπόν αυτούς τους στόχους ανάπτυξης των δραστηριοτήτων των τοπικών αλιών. Αυτά ε, ήθελα να πω. Ούτως ή άλλως συστηματικά σας αποστέλουμε όλα τα σχετικά έγγραφα και βεβαίως μπορούν μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, που θέλουν να παρακολουθήσουν τις εργασίες των ε, μικτών επιτροπών είναι καλόδευτη. Νομίζω ότι θα είναι επωφελής για όλους μας. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε Αλεξάνδρου. Δίνω και πάλι το λόγο στον εισηγητή για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση αυτό το θέμα. Κύριε Καντέκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Ζωζέφα για την παρέμβασή της. Επίσης, θα ήθελα να δείτε τι ωραία γραβάτα φοράει ο πρόεδρος, με τόνους. Σας ευχαριστώ κύριε Αλεξάνδρου για τις απαντήσεις σας. Ένα θέμα που έθεσε η Ιζαμπέλα δεν απαντήσατε. Τα παραλίευματα. Έχετε να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες. Περιμένει η Ιζαμπέλα την απάντηση. Ναι, κύριε Ισηγητά. Το ξέχασα, κύριε Πρόεδρε. Όπως ξέρετε, στη συμφωνία με τις Σεϊχέλες γίνεται στα πλαίσια των συμφωνιών για τα τονοειδή του Ινδικού ωκεανού. Και εμείς σε διμερές επίπεδο ακολουθούμε τις συστάσεις που έχουν εκδώσει η, η ΣΕΠΕΟΗ, η Επιτροπή Τόνου του Ινδικού Ωκεανού. Ό,τι λοιπόν κάνει επηρεάζει άμεσα ε, και απευθείας τις ε, διμερείς δικές μας ε, συστάσεις. Έχετε πληροφορίες για νέες δραστηριότητες πειρατείας που αφορά κοινοτικά αλλιευτικά ε, σκάφη. Δεν έχουμε τίποτα καινούργια προσέσουμε προσθέσουμε προς το παρόν. Αλλά βεβαίως δεν έχουμε καμία εγγύηση ότι στο μέλλον δεν θα υπάρξουν γεγονότα που θα επηρεάσουν αρνητικά το αλλιευτικό μας στόλο. Στο παρελθόν ξέρουμε ότι υπήρξαν επιθέσεις ε, πειρατών σε πολλά αλλιευτικά σκάφη που αλλιεύουν τόνο και κάποια από αυτά τα αλλιευτικά σκάφη ε, ακινητοποιήθηκαν, εκ των υστέρων απελευθερώθηκαν, αλλά τώρα τελευταία πρέπει να πω ότι δεν έχουμε πληροφορίες για αλληλευτικά σκάφη κοινοτικά τα οποία να έχουν ακινητοποιήσει οι πειρατές. Όταν, ε, κύριε Αλεξάνδρου, ε, είπατε ότι έγιναν ε, προσπάθειες για να απελευθερωθούν τι εννοείτε, πώς απελευθερώνονται, καταβάλλονται λίτρα ή με... Διότι πώς ελευθερώνεστε, ή καταβάλλετε λίτρα ή ε, αναπτύσσετε μια στρατιωτική δραστηριότητα. Τι εννοείτε εσείς, τι, πώς απελευθερώνονται αυτά τα αλληλευτικά σκάφη. Είναι απλή απάντηση. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε η Επιτροπή καταβάλουν λίτρα. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Καντέκ, σε σχέση με την πειρατεία, νομίζω θα πρέπει να είμαστε ε, σαφής. Απ' τη μια υπάρχει η επιχείρηση Αταλάντη και απ' την άλλη, δεδομένου ότι πρόκειται κυρίως για λιευτικά σκάφη ε, γαλλικά και ισπανικά. Στα γαλλικά αλευτικά σκάφη υπάρχει πάντα κάποιος από την ε, στρατιωτικός και το ίδιο συμβαίνει με το προσωπικό ασφαλεία στα ισπανικά. τα λιευτικά αυτά σκάφη, οι τράτες αυτές με τα παραγάδια από τη στιγμή που τα κλείνουν ε, μπορούν να αποχωρήσουν, αλλά εκείνη τη στιγμή είναι ευάλωτο. Τώρα όσον αφορά κάποια ρήτρα έχουν ήδη καταβληθεί, φαντάζομαι οι ίδιοι εφοπλιστές ή τα κράτη. Τώρα για να επανέλθουμε στην έκθεση. Σας ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας. Μπορείτε, αν δεν σας ικανοποιεί το περιεχόμενο της έκθεσης, βέβαια να καταθέσετε τροπολογίες. Προθεσμία κατάθεση τροπολογιών 27 Απριλίου το μεσημέρι. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, λοιπόν, αν θέλετε να καταθέσετε τροπολογίες, είστε ελεύθεροι. Βεβαίω, πρόκειται για ε, γνωμοδότηση, πρόκειται για γνωμοδότηση. Κανένα όμω δεν εμποδίζει. Κανένα να καταθέσει τροπολογίε. Α, πολύ περιορισμένε πρέπει να είναι, μου λέει ο γραμματέα. Λίγε, λίγε. Και αν δεν καταθέσετε και καμία, ακόμη καλύτερα. Ευχαριστώ κύριε Καντέκ. Όντω η προθεσμία είναι 27 Απριλίου το μεσημέρι. Και να διευκρινίσω ότι εδώ εμπίπτουμε στην ε, πλαίσιο της, ε, του, του άρθρου 218 της ε, Σέγγιν Λισαβόνας, ε, ότι δηλαδή οι τροπολογίες στο, στο κείμενο δεν μπορεί να είναι διαφορετικές, δεν μπορεί να είναι πολλές παρά περιορισμένες θα πρέπει λοιπόν όλοι να γνωρίζουμε αυτό το άρθρο 2.18 της Εθνικής Λισαβόνας ε, ότι θα μας βοηθήσει στις εργασίες μας. Ευχαριστώ, όπως είπα και στην αρχή, η κυρία Γιώτοβα δεν θα φτάσει στη συνεδρίαση παρά μετά τις 10.30. Θα ήταν δυνατόν τώρα να περάσουμε στο σημείο 7 της μεσαίας διατάξεως. Κλείνει το μικρόφωνο του Πρόεδρου. Είναι το έκθεση του κυρίου Κάπουλα Σάντο πρόκειται για το νέο πρωτόκολλο σχετικά με τον καθορισμό αλληλευτικών δυνατοτήτων και τη χρηματική αλληλεπαροχή που τη συμφωνία αλληλευτική σύμπραξη μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τη Λαϊκή Δημοκρατία του ΣΑΤΟΜΕ και Πρίντσιπε. Η πρόταση τη Κομισιόν βασίζεται στο άρθρο 43.2 σε συνδυασμό με το άρθρο 218 της συνθήκης της Λισαβόνας ε, επαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου. Οι σοσιαλιστές ανέλαβαν ε, την κατάρτιση της εκθέσεως και ο κ. Κάπουλα ορίστηκε εισηγητής ε, Στη συνεδρίασή μα τη 1η Φεβρουαρίου η Κομισιόν μα εξήγησε το περιεχόμενο τη προτάσεω και σήμερα ο κύριο ε, Κάπουλα ε, θα παρουσιάσει το σχέδιο γνωμοδότηση. Σχέδιο ε, σύσταση, συγγνώμη. Παρακαλώ, κύριε Σιγητά, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αρχίζοντα θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη διότι έφτασα με καθυστέρηση. Δυστυχώ όμω. Όπως ξέρετε είμαι συντονιστής ε, της πολιτικής μου ομάδας στην ε, Γεωργία και συστηματικά υπάρχει επικάλυψη των εργασιών αυτών των δύο επιτροπών. Είναι κρίμα, διότι έχουμε να κάνουμε με δύο ε, θέματα συναφή και σχεδόν οι ίδιοι βουλευτές παρακολουθούν αυτές τις δύο δραστηριότητες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όποιος θέλει να είναι παρόν και στις δύο επιτροπές έχει τρομερές δυσκολίες. Όπως είπε ο Πρόεδρος, πρόκειται για σχέδιο Σύστα σχετικά με την πρώτη απόφαση συμβουλή τη Σύνεψη Νέου Πρωτοκόλλου μεταξύ Ευρωπαϊκή Κοινότητα Λαϊκή Δημοκρατία Σάουτο και Πρίνσιπε. Το Σάουτο και Πρίνσιπε είναι μια ε, πρώην πορτογαλική απικία, παραδεισιακά νησιά, εξαιρετικά ωραία νησιά. Αν μπορέσετε να κάνετε εκεί διακοπές θα σας ε, ε, ενθουσιάσουν. Η μία βρίσκεται κοντά στον Ισημερινό ε, και η άλλη είναι πραγματικά και το μέρος στο οποίο αναπτύσσονται οι δραστηριότητες ενός εξαιρετικού βιβλίου ενός Πορτογάλου συγγραφέα που λέγεται Εκουαδόρ, σημερινός. Πρόκειται λοιπόν για εξαιρετικά ωραία νησιά. Έχουμε να κάνουμε με την ε, νέα συμφωνία με αυτά τα νησιά. Έξι μήνες μετά από την λήξη του πρώτου, συμφωνίας του πρώτου πρωτοκόλου ε, η Κομισιόν λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα. Έχουν ε, λοιπόν προσωρινά παραλύσει δραστηριότητε για τη συμφωνία αυτή. Πρόκειται για μία συμφωνία στα πλαίσια συμφωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, με τρίτες χώρες. Η ετήσια χρηματική αντιπαροχή είναι 682.500 ε, ευρώ υπάρχει ένα ετήσιο ποσό το οποίο ε, αυξήθηκε σε ύψος 455.000 ευρώ για την αποκλειστική οικονομική ζώνη Σαοτομέ και Πρίνσιπη. Έχουμε να κάνουμε ε, με ποσότητα αναφορά 7.000 τόνους ετησίως. Ε, σύμφωνα με τις διάφορες μελέτες επιπτώσεων έχει ε, αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει πρόβλημα υφορία για όλα τα είδη τόνου που αλλιεύονται, που είναι το κύριο ε, αλλιεύμα της περιοχής, έχει να αυξηθεί ε, λίγο αριθμό των σκαφών που αλλιεύουν, γρηγρή και παραγαδιών. Είχαμε περίπου σε ποσοστό 60-40 με τράτες γρηγρή και παραγάδια. Και οι ποσότητες ε, ε, αναφοράς μέχρι το 2010 ήταν 8.500 τόνοι ετησίως. Η όλη θεώρηση για το πρωτόκολλο αυτό είναι θετική. Αναγνωρίζει ότι έγιναν ε, πολλά θετικά εκ μέρους των αρχών του ΣΑΟ, των ΜΕ και Πρίνσιπε για τη Νέα Συμφωνία. Υπάρχει παρακολούθηση μέσω δορυφόρου, με την ε, βοήθεια των ε, οργανώσεων αλλιευάτων για τον ε, τόνο ε, υπάρχει βελτίωση. Η Μικτή Επιτροπή συνεδρίασε μία μόνο φορά. Δεν ξέρω πώς έκανε μία τέτοιου είδους ε, ε λεπτομερή ε, εξέταση του όλου θέματος με μία μόνο συνεδρία. Θα ήθελα εγώ να σας πω ποιο είναι το πρόβλημα το οποίο αντιμετώπισα και διαμαρτύρομαι έντονα. Ποιες είναι, ποιοι είναι οι κανόνες που ισχύουν για την διαβούλευση με τους βουλευτές που ασχολούνται με τα θέματα αυτά. Νομίζω ότι πρόκειται για θέματα τα οποία πραγματικά είναι ε, πάρα πολύ δύσκολα. Τι σημαίνει αυτό, ότι εγώ θα πρέπει να στείλω έναν υπάλληλο στην Επιτροπή να παρακολουθήσει την όλη υπόθεση. Ε, πραγματικά ένα μυστήριο επικρατεί για έγγραφα τα οποία δεν έχουν τίποτε το απόρριτο. Φαντάζεστε εάν πρέπει κάποιος να πάει, αν θέλει να δει και αν πρόκειται για τον ίδιο τον επίτροπο για κάποιον άλλο, αν θέλει πραγματικά να εξετάσει ένα έγγραφο, πρέπει να το κάνει με τι συνθήκες ασφαλείας, παρουσία ενός αξιωματούχου. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ατιμωτικό. Τι γίνεται δηλαδή. Και εγώ πρέπει να σας πω ότι εμένα πάντα με ελέγχαν οι υπάλληλοι. Δεν λέω ότι δεν ήταν συμπαθείς και ευγενείς και η παρέα τους ήταν εξαιρετική. Αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι αυτό είναι απαράδεκτο. Είναι ατιμωτικό αυτό το γεγονός. Δεν μπορούμε ε, εμείς στο κοινοβούλιο να υφιστάμεθα τέτοιου είδους ελέγχους. Εν πάση περιπτώσει Πρέπει να σας πω ότι η συμφωνία είναι σωστή, σταθμισμένη βεβαίως, υπάρχουν και διάφορες ρήτρε οι οποίες προβλέπουν την ε, ε, αναστολή των δραστηριοτήτων και την εφαρμογή του πρωτοκόλου σε κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις, αν υπάρχει παραβίωση στοιχείων ανθρωπίνων δικαιωμάτων κτλ. όπως προβλέπονται από τις συμφωνίες. Αλλά νομίζω ότι στην ε, συγκεκριμένη περίπτωση και για την Αφρική μπορούμε να θεωρήσουμε ότι λειτουργούν οι χώρες αυτές με τρόπο δημοκρατικό. Είναι σημαντική αυτή η συμφωνία και για το Σάτομα και Πρίσιπη και κυρίως για την ε, ε, κοινοτική αλληλεία στην περιοχή ε, μιλήσαμε προηγουμένως για την ασφάλεια στο Δυτικό Ινδικό, τώρα μιλάμε για ασφάλεια στον Ατλαντικό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή εκ των προτέρων, διότι έγκαιρα θα πρέπει να αποστέλει όλες τις πληροφορίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και επαναλαμβάνω ότι θα θέλαμε να έχουμε παρατηρητές στις μικτές επιτροπές και είμαστε πάντα στη διάθεσή σας αλλά υπό συνθήκε που δεν θέτουν σε αμφισβήτηση την αξιοπρέπειά μα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, συνάδελφοι. Ευχαριστώ για την εργασία σα επί τη εκθέσεω, κύριε Κάπουλας. Συμφωνώ απόλυτα ε, σε αυτά που είπα σχετικά με την αξιοπρέπεια των μελών. Πρέπει λοιπόν να το ξαναδούμε το ζήτημα. Το θέμα έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο ε, εξετάζουμε τις υποθέσεις ε, εταιρικών σχέσεων, συμπράξεων κλπ. Εντάξει, εμείς ε, έχουμε παρατηρητές στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων αυτών των συμφωνιών. Γιατί όμως υπάρχουν αυτά τα προβλήματα να θέλουμε να δούμε κάποια έγγραφα, γιατί μας μεταχειρίζονται με τον τρόπο με τον οποίο ανέφερε ο κύριος ε, Κάπουλας. Ε, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να υπομένουμε μια παρόμοια κατάσταση. Κυρία Λάβλεν. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και ε, σας κύριε Κάπουλα Σάντος για την έκθεσή τους. Ήμουν ε, γνωμοδότη, μάλλον συνέταξε γνωμοδότηση από την ε, αρμόδια επιτροπή, στην Επιτροπή δηλαδή Ανάπτυξης και πολύ ευχαρίστω να ξαναθέσω τα ερωτήματα που είχα θέσει τότε. Το βασικό και θεμελιώδης ζήτημα των, της συνεδρίασης ε, της, ε, της Επιτροπής, η οποία συνεδρίασε άπαξ και διερωτώ τι νέες ε, διατάξεις προβλέπει η Κομισιόν προκειμένου αυτή τη φορά να υπάρξουν συνεδριάσεις ε, της, ε, της Επιτροπής. Τώρα, ό,τι φορά την αξιολόγηση, δεν υπήρξαν παρατηρητές ε, επί των σκαφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόνο ότι αυτό προβλέπεται από τη Συμφωνία και απαιτείται. Τι νέες διατάξεις λοιπόν η Κομισιόν προβλέπει να θέση ώστε να υπάρχουν ε, επί των ε, αλληλευτικών σκαφών παρατηρητές Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε τώρα με τα αλλιεύματα δεν κατέτει σαφές πόσο αλλίευσαν τα σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πώς θα λαμβάνουμε τα πραγματικά στοιχεία αυτή τη φορά συμπεριλαμβανομένου και των παραλλιευμάτων. Ε, Επίση, των τόνο αλλά και τους καρχαρίες και τις θαλάσσιες χελώνες. Στη γνωμοδότησή μου επίσης ε, αναφέρω πως ε, σύμφωνα με την αξιολόγηση υπήρξαν σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δραστηριοποιούνταν στην περιοχή αλλά έφεραν σημαία άλλου κράτους. Ε, λοιπόν, η Κομισιόν πώς θα πρέπει να ε, μπορεί να ελέγχει ότι τα σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα πρέπει να φέρουν αλεύοντας στην περιοχή σημαία άλλου κράτους. Και τέλος ε, να συμφωνήσω απόλυτα με τον Κάπουλα Σάντος αναφορικά με τις εκθέσεις αξιολόγησης και την όλη διαδικασία που θα ακολουθεί προκειμένου να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας ε, ως ε, εκλεγμένοι εκπρόσωποι των ε, Ευρωπαίων πολιτών. Θα πρέπει λοιπόν να μπορούμε να έχουμε όλα αυτά τα έγγραφα που φορούν στις αξιολογήσεις διάθεσή μας πληρώνονται στο κάτω-κάτω με χρήματα των φορολογουμένων και εμείς είμαστε άμεσα εκλεγμένοι από τους Ευρωπαίους πολίτες και πρέπει να έχουμε τα χέρια μας σε αυτές τις αξιολογήσεις ε, προκειμένου να έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε τη δουλειά μας σωστά και απροβληματικά ε, το όνομα της διαφάνειας. Ε, αυτά ήταν τα σχόλιά μου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Μία σειρά ακόμα ερωτήσεων προς τον κύριο Αλεξάνδρου από την DG μάρα Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στα ερωτήματα της κυρίας Λόβιν που ήταν ε, πολύ καλά στοχευμένα, που φαίνεται πως ε, ελέγχει απόλυτα και με μπρίο το περιεχόμενο όλων αυτών των πρωτοκόλων αναφορικά με την διαδικασία. Κάθε φορά που έρχομαι στο Κοινοβούλιο ακούω παράπονα για το ότι αυτές οι εκθέσεις ε, αξιολόγησης ex post φτάνουν στο Κοινοβούλιο με, τον, με τη σφραγίδα εμπιστευτικό έγραφο, αλλά αυτό δεν είναι κάτι το οποίο εγώ μπορώ να αλλάξω. Κάθε φορά ακούω τα παράπονα, τα αναφέρω στους αρμοδίους, αλλά όπως καταλαβαίνετε δεν είναι ένα ζήτημα που εμπίπτει στις αρμοδιότητες μου και στις δυνατότητες μου. Ε, δεύτερο σημείο το γεγονό ότι το προηγούμενο πρωτόκολλο με το ΣΑΟ Τόμε δεν ε, έγινε παρά μόνο μία συνεδρία της Μικτής Επιτροπής και θα πιστεύετε ότι μία και μόνο συνεδρίαση δεν επιτρέπει την παρακολούθηση της ε, εφαρμογής του πρωτοκόλλου. Συμφωνώ μαζί σας, δεν είναι και μοναδική περίπτωση, το διαπιστώσαμε και στον Ειρηνικό, η κυρία είχε τονίσει αυτήν την ε, αδυναμία. Με ρωτάτε ποια είναι τα μέσα τα οποία έχουμε στο παράρτημα προκειμένου να τηρηθεί η συμφωνία. Δεν έχει κανένα συμπληρωματικό μέσο. Προβλέπεται το παράρτημα μια ε, συνεδρίαση κατέτος και είπα και ξανάπα, γιατί είναι μια προσωπική μου δέσμευση, ότι φροντίζω τι υποχρεώσει ε, να τις στηρούν και οι μεν και οι δε και οι δύο πλευρές. Ε, γι' αυτό λοιπόν προσπαθούμε να συγκαλούμε συνεδριάσεις μικτών επιτροπών για όλα τα πρωτόκολλα. Τελευταίου 15 μήνες συγκαλέσαμε 14 ή 15 μικρές ε, επιτροπές. Είναι τεράστια η 15 μεικτε επιτροπε ειναι σχέση με το παρελθόν, αλλά όπως καταλαβαίνετε έχουμε περιορισμένους ε, ανθρώπινους πόρους και δεν μπορούμε ταυτόχρονα να καλύπτουμε τα πάντα. Αλλά έχουμε τη θέληση και έχουμε την πρόθεση να τηρήσουμε αυτήν την ε, δέσμευση, την υποχρέωση που είναι ε, πρωταρχική σημασία, όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για την τρίτη χώρα. Να έχουμε αυτήν την κοινή την, την συνάντηση με στο πλαίσιο της Επιτροπή. Τώρα, δεν υπάρχει υποχρέωση στο πρωτόκολλο με το ΣΑΟ ΤΟΜΕ αναφορικά με την ε, ε χρησιμοποίηση παρατηρητών. Ε, υπάρχουν διαδικασίες σχετικά με την ε, χρήση παρατηρητών επί των σκαφών. Είχαμε πει ότι θα πρέπει να φροντίσουν πως αν υπάρχει έλλειψη παρατηρητών να φροντίσουν ώστε να εξευρεθούν και να εκπαιδευτούν νέοι παρατηρητές ώστε να είναι στη διάθεση των αλληλευτικών στολίσκων που αλλιεύουν στην ΑΟΖ του Σαοτόμε. Όταν λοιπόν ε, θα ξανασυναντήσουμε τους ε, Σαοτομανούς θα τους ζητήσουμε να προβλεφθεί δράση για την εκπαίδευση προσωπικού, διότι συχνά μας λένε ότι δεν έχουν τεπιμένο προσωπικό. Εάν έτσι έχουν τα πράγματα, τότε πρέπει να προωθήσουν την εκπαίδευση παρατηρητών ε, όπου προβλέπετε, από την κλαδική στήριξη. Τώρα σε φορά τα αλλιεύματα έχουμε μια διαδικασία που ε, προβλέπεται στο παράρτημα για τη δήλωση των αλλιευμάτων. Αυτές οι δηλώσεις ε, ε, επικυρώνονται από τις επιστημονικές οργανώσεις τις ευρωπαϊκές, δεν πρόκειται για την ΕΟ, για τον Ισπανικό στολίσκο ή την ERD για τον Γαλλικό στολίσκο. Ε, δεν βλέπω για ποιο λόγο υπάρχει πρόβλημα εδώ των αντίον ε, η παρατήρηση που έγινε αναφορικά με τις ε, σημαίες ευκαιρίες και το ε, θέμα της αποκλειστικότητας. Ξέρετε ότι έχουμε σε όλες τις συμφωνίες ρήτρα αποκλειστικότητας και επιθυμούμε αυτή η ρήτρα να τηρείται και από τους και από δε. Παρατηρήσαμε ότι υπάρχουν κάποια σκάφη που αλλάζουν σημαία, το ονομαζόμενο reflagging, αλλάζουν επισύοντα. Λοιπόν, το έχουμε προβλέψει για το μέλλον στο πλαίσιο της ε, άσκησης για τη μεταρρύθμιση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής, ειδικά η επιτυχή που αφορά στην εξωτερική δράση, έχουμε προβλέψει ε, την ε, δυνατότητα για την καταπολέμηση του reflagging της αλλαγής επισύοντα. είναι πολύ νωρίς να σας πω τις λεπτομέρειες, βρίσκεται στα σκαριά το ζήτημα θα λάβετε όμως μία ανακοίνωση και στην ανακοίνωση αυτή θα δείτε πως υπάρχει ένα σημείο σχετικά με το reflagging και εμείς κρίναμε ότι έρευε να αντιδράσουμε προκειμένου να μην διακινδυνεύσουμε την ρήτρα αποκλειστικότητα και να διασφαλίσουμε ισότιμη μεταχείριση όλων των Ευρωπαίων εφοπλιστών όταν αλλιεύουν σε αυτές τις ε, αποκριστικές ζώνες. Ευχαριστώ κύριε Αλεξάνδρου. Θέλετε να ολοκλώσετε τη συζήτηση κύριε Κάπουλης. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή για τις διευκρινήσεις και την κυρία Λόβιν για τις ε, διευκρινήσεις της όσον αφορά το τελευταίο θέμα που αφορά. Θα ήθελα να πω ότι αλλιεύουν αλλιευτικά σκάφη τρίτων χωρών ε, στην περιοχή σάτομε και Πρίνσιπε, Ιαπωνικά, από την Ταϊβάν. Δεν γνωρίζουμε τον ακριβή αριθμό. Απλώς θα ήθελα ε, να διευκρινιστεί περαιτέρω το θέμα αυτό. Αν μπορεί να έχει πιο συγκεκριμένα στοιχεία μας παρουσιάσει η Επιτροπή. Ε, κατά τα άλλα πρέπει να πω ότι εγώ είμαι στην διάθεση όλων για να μπορέσει να ολοκληρωθεί η έκθεση και θα ευχαριστώ τους συναδέλφους που θα θελήσουν να καταθέσουν τροπολογίες σχετικά. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κάπουλα Σάντος. Κάνατε μια πολύ καλή δουλειά και για το Σαρωτομεγία του Ε, Προθεσμία για τη διάθεση τροπολογιών είναι 27 Απριλίου το μεσημέρι, όπως ε, και με την προηγούμενη έκθεση που εξετάσαμε. Και να επενθυμίσω στα μέλη ότι αυτό ε, εξετάζεται σύμφωνα με το άρθρο 218 6α, ότι δηλαδή θα πρέπει να απαντηθεί ναι ή όχι στην, ε, και μόνο τεχνικής φύσης τροπολογίες θα πρέπει να εξεταστούν. Σας παραλαμβάνω ότι δεν έχουμε ε, λάβει κάποιο έργο από το Συμβούλιο, την ανάθεση από το Συμβούλιο, γι' αυτό δεν θα υπάρξει, ε, δεν ξέρουν πότε θα, δεν ξέρουν πότε θα ψηφιστεί το, το θέμα από την Ολομέλεια. Μέχρι ότου λοιπόν ε, συμβεί αυτό, δηλαδή λάβουμε την ανάθεση, τότε μέχρι τότε δεν μπορούμε να... Δεν μπορώ μάλλον να σας πω περισσότερο. Χαίρομαι που η κυρία Ιώτοβα ήρθε ανάμεσά μας ε, και θα εξετάσουμε το θέμα σας που είναι το υπαρθμόν 6 και θα ενθυμίσετε ότι την 18η Μαΐου πέρυσι οι συντονιστές αποφάσισαν να υπάρξει μια έκθεση πρωτοβουλία για την τρέχουσα και μελλοντική διαχείριση της αλίας στον Εύξηνο Πόντο και να θέσω στην κυρία Ελιάνα Μαλίνοβα να αναλάβει την έκθεση. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που κάνετε αυτή την αλλαγή στη μέσα διάταξη, διότι στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ συζητήθηκε το θέμα της ένταξης ε, της ε, Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Συμφωνία Σέγγεν. Σε ό,τι φορά την έκθεση για την τον έξινο πόντο, λάβατε το κείμενο και σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον που δείξατε. και στην ε, θέση που μας ε, ανέφεραν οι εμπειρογνώμονες που συναντήσαμε την περασμένη φορά. Νομίζω πως όλες οι προφορίες όσες θα λάβατε μέχρι τώρα θα σας ε, ενημερώνουν για το πρόβλημα και για τις προκλήσεις που υπάρχουν στον έξινο πόντο. Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις προφορίες που έλαβα μετά από τις επαφές που είχα με τις παράκτες αρχές περιοχές και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εκπροσώπους της DGMAR για την ε, πολύ καλή αντιμετώπιση να ευχαριστήσω επίσης και την Επίτροπο κυρία Δαμανάκη η οποία ανέλαβε να ξεκινήσει και να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις με όλους τους εμπλεκόμενους ε, της πυραβάνομης της Τουρκίας και της Ρωσίας. Πιστεύω ότι με την, ε, με την ε, δημιουργία μιας ρυθμισμένης κατάστασης ε, στην ε, περιοχή θα μπορέσουμε να επωφεληθούμε όλοι μας ε, διότι μέχρι τώρα η νομοθεσία είχε πάρα πολλές ελλείψεις είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία με τον κύριο Τσουκαλά ο οποίος δεν μπόρεσε σήμερα να παρευρεθεί στην συνεδρίασή μας και θεωρώ ότι μπορούμε να υποστηρίξουμε την άποψή του ότι δηλαδή όλες οι αποφάσεις που αφορούν τον έξινο τόμπο θα πρέπει να στηρίζονται σε επιστημονικές ε, μελέτες ε, και συμφωνίες ε, που θα έχουν γίνει μεταξύ των έξι παράκτιων κρατών. Ε, ακούσαμε επίση και τις θέσεις των συναδέλφων. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ρόγκουστ και την κυρία Αντρέα Μπαρέφ για την υποστήριξή τους. Δήλωσαν ότι χρειαζόμαστε ένα, πολύ σωστή και αποτελεσματική διαχείριση των ε, αλευτικών πόρων στην, στον ε, εύξηνο πόλο. Επίσης ε, να πούμε ότι ο συντονισμός των θαλάσσιων δραστηριοτήτων είναι πάρα πολύ σημαντικός. <clears throat> Θέλουμε να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα των αλληλευτικών πόρων και άρα την ε, χρησιμότητα των αλλίων μας και των αλληλευτικών μας τολίσκων. Χρειάζεται να λάβουμε επίσης ε, υπόψη την κατάσταση που επικρατεί σε όλες τις παράκτητες περιοχές. Να ευχαριστήσω την κυρία Λοβίν, η οποία ρώτησε πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν ακόμα αλληλευτικά αποθέματα στην ε, περιοχή αυτή, σε αυτήν την κλειστή λεκάνη. Ε, χρειάζεται να υπάρξει συνεργασία με διάλογος με τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τα άλλα κράτη που είναι παράκτια στον εύξηνο πόντο για να διασφαλίσουμε και την επιβίωση των ε, αλληλών μας. Ποιες είναι οι προκλήσεις λοιπόν που αντιμετωπίζουν στην ε, με την πόντο. Πρώτα απ' όλα, θεωρώ ότι μια καλύτερη διοικητική συνεργασία στον έξινο πόντο είναι κάτι το οποίο θα αποβεί προς όφελος όλων των παρακτών κρατών. Μέχρι τώρα δεν έχουν υπάρξει συμφωνίες. Επίσης χρειάζεται να εξτάσουμε το ζήτημα της χρηματοδότησης Παράλληλα, πρέπει να υπάρξουν πολιετή προγράμματα τα οποία θα αντικαταστήσουν ε, τα υφιστάμενα το υφιστάμενο σύστημα των ποσοστώσεων και οι οργανώσεις των αλλιέων θα πρέπει να δραστηριοποιηθούν περαιτέρω. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δώσουμε στην ε, αλλία μικρής κλίμακας <clears throat> να λάβουμε μέτρα για να εξαλείψουμε την παράνομη λαθρέα και αναρχή αλία. Και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι έχουμε εγκαίρως εγκρίνει την ε, έκθεση σχετικά με την πλά και με τον αθέμητο ανταγωνισμό ο οποίος ε, υπάρχει συχνά ανάμεσα στις παράκτιες χώρες. Τέλος, θα ήθελα να συμμεριστώ την άποψή ότι χρειάζεται να υπάρξει και η εμπλοκή ενό άλλου διεθνού οργανισμού στι δραστηριότητε του εύξηνου πόλου, διότι διαφορετικέ επιστημονικέ πληροφορίε που λαμβάνουμε δεν οδηγούν σε κάποια συμπεράσματα ακριβή. Γι' αυτό θα ήθελα να σας υπενθυμίσω πως ε, σύμφωνα με το προσωρινό χρονοδιάγραμμα η ε, κατάθεση τροπολογιών είναι 27 Απριλίου. Ευχαριστώ κυρία Γιώτοβα. Ε, θα ήθελα να μας απαντήσετε σε αυτό το ερώτημα για τα αλλιεύματα στη Μαύρη Θάλασσα. Κυρία Λόβεν, ε, ήταν ένα σοβαρό ερώτημα. Μου έκανε πάρα πολύ έντονη εντύπωση όταν ήρθα εδώ και είδα ότι δεν υπάρχει κανένα διαχειριστικό σώμα για την ε, ε, κατάρτιση ποσοστώσεων στην Μαύρη θάλασσα. Τέτοια προβλήματα ανάλογα είχαμε και στην ε, Βαλτική θάλασσα όπου η κατάσταση δεν είναι πάρα πολύ καλή αλλά οπωσδήποτε βελτιώνεται. Χρειάζεται απαραίτητο μια χρηστότερη διαχείριση. Πρέπει να υπάρχει ένα διαχειριστικό σώμα για τη Μαύρη θάλασσα και πιστεύουμε ότι αν υπάρξει θα πρέπει να το πλαισιώσουμε και να το υποστηρίξουμε. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να αναλάβει αυτή την πρωτοβουλία και να καταβάλει προσπάθειες για να συλλέξει όλα τα δεδομένα και να πάρει μαζί της όλες τις παράκτιες χώρες, ε, τα παράκτια κράτη της Βόρειας Θάλασσας, ε, γιατί είναι και αυτή πλέον μια ευρωπαϊκή θάλασσα. Διαβάσαμε την εκθεσή και συμμεριζόμαστε το περιεχόμενο του σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έχω ορισμένα ερωτήματα. Το πρώτο αφορά, υποθέτω ότι η κυρία θεωρεί ότι στην έκθεση λέει ότι θα πρέπει να υπάρχουν ε, ποσοστά για τους ε, Βούλγαρους και Ρουμάνους αλλής, ε, θα πρέπει να υπάρξει ένας ε, περιορισμός των ε, δραστηριοτήτων μακροπρόθεσμα, φαντάζομαι ότι αυτό εννοεί. Επίσης υπάρχει το πρόβλημα το An alien species and... του Βέιν το οποίο έχει μία ένα θαλάσσιο, ιαπωνικό θαλάσσιο σαλιγκάρι ε, χαρακτηριστικός θηρευτής ε, και λέγεται ραπάνα βενόσα. Χρειάζεται λοιπόν να προστατευθεί αυτό το, αυτή η ραπάνα βενόσα από τα άλλα αλλιεύματα τα οποία παραβλάπτουν ε, όλα τα ε, οστρακοειδή και όλον τον πληθυσμό των οστρακοειδών χρειάζεται να δώσουμε την δυνατότητα για τα αποθέματα γάβρου και παπαλίνας τα οποία έχουν αρχίσει να ανακάπτουν μέχρι ενό σημείο, βλέπουμε ότι πρέπει να προστατευτούν εν πάση περιπτώσει και ίσως θα μπορούσατε να μας εξηγήσετε την ιδέα που στηρίζει αυτά η κυρία Γιώτοβα μπορεί να μας πει πώς θα ξαναυπάρξει, ε, θα ανακάμψουν τα λιεύματα και θα ξαναυπάρξει αλία. Ε, τα ερωτήματά μου είναι αυτά και τώρα θα ήθελα να σας ευχηθώ καλή τύχη πραγματικά γιατί είναι μια πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία η έκθεση αυτή. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να ζητήσω από την κυρία Άντας Μαρίνα Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κυρία Γιώτοβα για την ε, παρουσίαση αυτής της ε, έκθεσης ε, που πραγματικά θέτει τον δάκτυλο από τον τύπο των ήλων για ένα ζήτημα πολύ σημαντικό διότι είναι ένα ουσιαστικό ζήτημα και αναφέρομαι στο συντονισμό ανάμεσα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με χώρες ε, μη μέλη τη Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα πρέπει να συνεργαστούν και να διευθετήσουν αυτό το πρόβλημα για την δημιουργία ενός οργανισμού για την διαχείριση της αλίας των έξων απόλυτων. Μιλάμε για την Ρωσία και την Τουρκία που είναι κράτη σημαντικά που θα πρέπει να ε, συνεισφέρουν ένα πρόγραμμα διαχείρισης μακροπρόθεσμο για τον καθορισμό του επέδου των αλλιευμάτων ε, και επίσης το ζήτημα της ε, βιωσιμότητας των παράκτων περιοχών και των αλλιών τους που ζουν αυτή τη δραστηριότητα. Κυρία Ιάτοβα μίλησε για την παράνομη αλλία. Είναι φυσικά ότι μάλλον είναι απαραίτητο να υπάρξει μια συνεργασία για να καταπολεμηθεί αυτή η παράνομη αλλία. Είπατε ότι χρειάζονται κονδύλια, χρειάζονται χρήματα μια περιοχή η οποία δεν έχει καμία ρύθμιση στον τομέα αυτό, είναι προφανές ότι χρειάζεται να υπάρξει, να δοθεί μια τάξη και να εξελιχθούν κάποια κονδύλια τα οποία θα διατεθούν. Ευχαριστώ κυρία Ιετοβά. Ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα τώρα να ζητήσω από την ε, Γενική Διευθυνσή Μάρε, τον κύριο Τωρατέρα, να μας απαντήσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελε η Επιτροπή να συμφωνήσει με τα συμπεράσματα της κυρίας Γιώτοβα να την ευχαριστήσει για την εξαιρετική συνεργασία κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας αυτής της εισήγησης. Πολύ συχνά συνεργαστήκαμε και συμβάλαμε από δικής μας πλευράς, από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οφείλω να πω ότι είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι, όχι μόνο για το αποτέλεσμα, αλλά και για την δυνατότητα η οποία μας δόθηκε να έχουμε ανταλλαγή όχι μόνο πληροφοριών, τις οποίες διαθέταμε και εμείς από δικής μας πλευράς, αλλά και ε, διάφορες πρωτοβουλίες ε, που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις οποίες προωθεί η κυρία Γιώτοβα, πρωτοβουλίες που έχουν σαν στόχο να τονίσουν την αναγκαιότητα ε, της ε, συντήρησης ε, των αλλιευμάτων στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Πολύ σύντομα πρέπει να πω ότι στα περισσότερα σημεία που θίγησαν σε αυτή την έκθεση κύριε Πρόεδρε υπάρχουν σημεία πάρα πολύ κρίσιμα για τη Μαύρη Θάλασσα και είμαστε σύμφωνοι με το περιεχόμενο αλλά και με τον τρόπο προσέγγισης τους. Δηλαδή ένα, υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης επιστημονικής συνεργασίας. Δύο, να υπάρξει μεγαλύτερη προσπάθεια, αύξηση της προσπαθίας με τις παράκτιες χώρες μαζί για να καταπολεμηθεί η παράνομη αλληλεία και επίσης ανάγκη να υπάρξει μια ολοκληρωμένη ε, θαλάσσια πολιτική για την ε, Μαύρη Θάλασσα. Αρχίσαμε ήδη να δουλεύουμε πάνω σε όλα αυτά τα σημεία και ο Επίτροπός μας ε, είναι ε, συμπράτη ε, και το ξέρει αυτό η κυρία Γιώτοβα. Είναι για μας πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά τα στοιχεία. Επίσης θα ήθελα να το βάλω ένα σχόλιο για το θέμα της διαχείρισης των πόρων και της ε, δυνατότητας να έχουμε μια συγκεκριμένη οργάνωση για την Μαύρη Θάλασσα, αλλά και για το θέμα των μεγίστων δυνατών αλλιευμάτων και των ποσοστώσεων. Το να ε, εγκριθούν μακροπρόθεσμα σχέδια διαχείρισης δεν είναι αντίθετο με ένα σύστημα τάκ και ποσοστώσεων και δηλαδή μεγίστων αλλιευτικών ποσοτήτων και ποσοστώσεων, και, αλλά εδώ υπάρχει μια δυσκολία. Η δυσκολία είναι στην εφαρμογή γιατί σήμερα δεν έχουμε ούτε ε, στο πλαίσιο της οργάνωσης που διασχίζει την ε, Μαύρη Θάλασσα και την Μεσόγειο, δεν έχουμε τη δυνατότητα να διαχειριστούμε από κοινού τα αλλιεύματα και τους πόρους κυρίως τους πόρους έχουμε αναλάβει μια σειρά αποδράσεις. Έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε έναν ειδικό οργανισμό, αλλά αυτό απορροφά και πόρους και χρόνο. Ε, επίσης πρέπει να πάρουν μέρος όλα τα φορόμενα μέρη και τα ενδιαφερόμενα μέρη. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι πολιτικά το θέμα πολλές φορές στην περιοχή αυτή. Το εγχείρημα αυτό ξεπερνά το πρόβλημα της αλίας και της θαλάσσιας ολοκληρωμένης πολιτικής βεβαίως. Είναι ένα στόχος ωστόσο τον οποίο μπορούμε να τον καθορίσουμε μακροπρόθεσμα, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να υπάρξει μια μέγιστη χρησιμοποίηση των οργανώσεων που υπάρχουν ήδη, που μας επιτρέπουν να προχωρήσουμε, ούτως ώστε να έχουμε έναν καλύτερο συντονισμό των πολιτικών και μεσοπρόθεσμα να έχουμε μια οργάνωση η οποία να αναλάβει την Μαύρη Θάλασσα και να συνεχίσει να μελετά μαζί με τα κράτη-μέλη και το Κοινοβούλιο αλλά και τις άλλες ε, παράκτιες γειτονικές χώρες. Αυτό το σχόλιο ήθελα να υποβάλω για να διευκρινίσω ότι από δική μας πλευρά συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με αυτά που υπάρχουν ήδη σήμερα ό,τι υπάρχει. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα υπάρχοντα εργαλεία για να έχουμε ένα καλύτερο συντονισμό των πολιτικών συντήρησης. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Ντοντέλα. Θα ήθελα απλώς να επαναλάβω αυτό που είπε η κυρία Λαβέν, κυρία Γιώτοβα. Εάν προτείνεται για τη Ρουμανία και την Βουλγαρία να έχουν ορισμένες ποσοστώσεις ε, στην θάλασσα και συσχετίζεται και με την Τουρκία και τις άλλες παράκτιες ε, χώρες, πώς θα οργανωθεί η αλίευση στην Μαύρη Θάλασσα. <coughs> Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα απαντήσω τις ε, ερωτήσεις των συναδέλφων μου τώρα. Υπάρχει ένας ρόλος που είναι που πρόκειται να αναλάβουμε, που είναι κοινό. Μερικά χρόνια πριν η, η Βουλγαρική Βουλή ενέκρινε ένα νόμο ο οποίος ρητά απαγορεύει την, ε, τον έλεγχο στις, ε, στη Μαύρη Θάλασσα. Αν διαβάσετε την αιτιολογική σκέψη αυτής της νομοθεσίας, βλέπετε ότι υπάρχει κάτι περίεργο. Υπάρχουν εμπορικά επιχειρήματα τα οποία υπερισχύουν των περιβαλλοντικών και δεν είναι μυστικό ότι υπάρχουν ε, πολλές πρώτες ύλες, ε, ε, ακριβές και ε, γίνεται εξαγωγή τους στην Ιαπωνία και σε άλλες χώρες. Βεβαίως ε, αυτό υπάρχει ως εμπορικό, εμπορική δικαιολογία, εμπορικό επιχείρημα. Αλλά μέσα στην Μαύρη Θάλασσα τα τελευταία χρόνια υπήρξε μεγάλη οικολογική καταστροφή και πάρα πολλά αλλιεύματα, πάρα πολλά είδη ηχθείων βρίσκονται σε κίνδυνο και πιστεύουμε ότι δεν θα έπρεπε να αφήσουμε ε, ελεύθερες αυτές τις δραστηριότητες. Θα πρέπει να υπάρξουν ορισμένες επιλογές. Θα πρέπει να γίνει μια επιστημολική ανάλυση με τα κατάλληλα συμπεράσματα και να λάβουμε ορισμένα προσωρινά μέτρα. Θα μπορούσε να είναι ένα προσωρινό μέτρο αυτό, η απαγόρευση ορισμένων δραστηριοτήτων. Λίγους μήνες πριν επισκέφτηκα τα αρμόδια σώματα, της αρμόδιες αρχές στην Άγκυρα και συζήτησα μαζί τους για το θέμα που έχει, όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την έκθεσή μου. Επίσης πρέπει να πω ότι έχουμε μία συμφωνία μεταξύ των κρατών της Μαύρης Θάλασσας τελικά θα καταλήξουμε σε μια εντελώς σταθμισμένη και ισορροπημένη έκθεση. Ε, στην ε, ε, Τουρκία όμως δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία και η Μαύρη Θάλασσα είναι μικρή, κλειστή και περιορισμένη. Θα έχουμε να τους εκπροσώπους της Τουρκίας με τους οποίους συμφωνήσαμε να αναθεωρήσουμε αυτή την νομοθεσία, να την εξετάσουν ε, ακόμα μία φορά, ούτω ώστε να μπορεί να υπάρξει μία κοινή βάση συνεργασίας σε ό,τι αφορά τα αποθέματα, τα αλλιευτικά στη Μαύρη Θάλασσα. Υπάρχει κάποια πρόοδος στην κατάσταση. Ε, θέσατε και άλλα ερωτήματα στην έκθεσή μου και στην παρουσίασή μου είπα πολλές φορές ότι ποτέ δεν υπήρξε μια κοινή συμφωνία μεταξύ των έξι παρακτήων κρατών της Μαύρης Θάλασσας. Και θα γίνω πιο άμεση και θα πω ότι μία από αυτές τις ε, έξι χώρες ε, η οποία ε, αλλιεύει στην ε, Μαύρη Θάλασσα βρά άναρχα και υπάρχουν συνέπειες για την Μαύρη Θάλασσα. Βουλγαρία και Ρουμανία είναι μέλη της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και σεβόμαστε τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι συστάσεις αυτές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν ισχύουν όμως για τις άλλες τέσσερις χώρες κατά κανέναν τρόπο. Ε, δηλαδή το 90% των αλλιευμάτων ε, δεν υφίσταται ούτε ποσόστος, ούτε περιορισμό, ούτε απαγόρευση ούτε τίποτε από όλα αυτά. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να ρυθμίσουμε τις σχέσεις μεταξύ των έξι, καταρχήν έξι παρακτήων χωρών και μετά σε σχέση με την κοινή αλλιευτική πολιτική στην οποία εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση όλοι είμαστε, ε, όλοι την προωθούμε. Πιστεύω επίσης γιατί μου έδωσαν διασφαλίσεις σε διάφορες συνεδριάσεις όπου ήρθα σε επαφή με Ρώσους συναδέλφους ότι υπάρχει κοινό έδαφος. Μπορούμε να βρούμε έναν τρόπο συνεργασίας αν είμαστε επικοδομητικοί και επαγγελματίες. Επίσης συζήτησα με εκπροσώπους ε, της Επιτροπής Μεσογειακής Αλίας και αυτή είναι η απάντησή μου. Βεβαίως μπορεί να υπάρξει ένα σώμα διαχειριστικό της ε, Μαύρης Θάλασσας. Αυτό γίνεται μια νυχτή. Αλλά πώς θα γίνει η εφαρμογή. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο θα πρέπει να μπορούμε να κάνουμε πλήρη χρήση των ευκαιριών που μας δίνει η Γενική Διεύθυνση ΜΑΡΕ. Ο στόχος μας είναι να μην έχουμε κυρώσεις ε, στην Μαύρη Θάλασσα με εμπειρογνώμονες οι οποίοι έρχονται στη Βουλγαρία και στην ε, Ρουμανία και οι οποίοι έχουν τις τύχες της αλίας στα χέρια τους. Θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν την κάθε δυνατή ευκαιρία που μπορεί να μας παράσχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εάν θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, καταρτήσει μια τέτοια οργάνωση η οποία ε, θα απορρέει από την Γενική Διευθύνση ΜΑΡΕ θα μπορέσουμε ίσως να προσπαθήσουμε να ε, παροτρύνουμε και τους άλλους να πάρουν μέρος Τελικά πιστεύω ότι υπάρχει και το θέμα της αγοράς των αλλιευμάτων. Πρέπει να ξέρουμε ότι χρειάζεται καταρχήν απολύτως η δέσμευση για την ισορροπημένη σχέση των έξι χωρών και μετά μπορούμε να περάσουμε στα επόμενα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Ήταν αυτό ένα πολύ θετικό συμπέρασμα. Έτσι φτάνουμε στο πέρας της συζητήσεως ε, της ε, έκθεσής σας. Ε, σας είμαι πάρα πολύ ευγνώμων που δαπανίσατε χρόνο και ενέργεια για τη σύνταξη αυτής της έκθεσης και νομίζω ότι τελικά θα καταλήξουμε στο να έχουμε μια κοινή συμφωνία με τις άλλες χώρες, τις έξι παράκτιες χώρες της Μαύρης Θάλασσας. Η προθεσμία καταθέσεων ε, για τις τροπολογίες την 27 Απριλίου επίσης. Τώρα ίσως θα μπορούσαμε να επανέλθουμε στην ημερήσια διάταξη και να περάσουμε στο θέμα 9 που είναι μια άλλη έκθεση πρωτοβουλίας ε, ε, για τον ρόλο της ΕΕ και την έκθεση της κυρίας Λόβεν η οποία είχε εγκριθεί στις 15 Σεπτεμβρίου από τη διάσκεψη των Προέδρων και η κυρία Λόβεν καθορίστηκε ως ε, η συγγήτρια. Η Επιτροπή Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος επίσης ζήτησαν ένα ε, σχέδιο έκθεση. Στις 27 Οκτωβρίου 2010 είχαμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων και της έκθεσης αυτής και στις 26 Ιανουαρίου του 2011 ε, η εισηγήτρια παρουσίασε το πρώτο έγγραφο εργασίας. Η κυρία Λόβεν σήμερα θα παρουσιάσει ένα δεύτερο έγγραφο εργασίας που ασχολείται με άλλες διεθνείς πρωτοβουλίες ε, ε, οι οποίες καλύπτουν την αλληλεία Αγιουγιού. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Λόβεν για το δεύτερο έγγραφο εργασίας και της δίνω το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτό είναι λοιπόν το δεύτερο έγγραφο εργασίας για, τον, ε, για την καταπολέμηση της παράνομης αλίας σε παγκόσμιο επίπεδο και το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να σας τονίσω το μέγεθος της, των προβλημάτων των ε, της, της ΕΕ. Υπάρχουν τεράστιες απώλειες χρηματοοικονομικές, πάνω από 10 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα στον τελευταίο χρόνο. 20% ε, των ε, αλλιευμάτων προέρχονται από την Αγιουγιού, κάτι το οποίο την καθιστά την πρώτη αλλιευτική δύναμη 16% των ποσοστώσεων επίσης μέσα στις, ε, στις ευρωπαϊκές θάλασσες ε, είναι της Αγίου και πιστεύουμε ότι πρέπει να τονίσουμε ότι η, η ρύθμιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαρτάται πλήρως από αυτό που αποκαλούμε ευθύνη για τις ε, κρατικές σημαίες. Ε, η πολλές φορές χρειάζεται ένα, κείμε, ένα εγγραφό που να πιστοποιεί ότι το τάδε αλίευμα ε, αλλιεύεται νομότυπα. Δεν υπάρχουν όμως τέτοια έγγραφα, ούτε μπορούν να παρασχεθούν. Για κάθε κράτος πρέπει να αναλυφθεί η ευθύνη ειδικά από το κράτος για την αλίευση, για τα ε, σκάφη και για, τα, για τους λιμένες. Πριν να παραχθεί η έκθεση είχε υπάρξει το πρώτο έγγραφο εργασίας που μιλούσε για τα μέτρα της καταπολέμησης της παράνομης αλίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Ε, καταρχήν σε παγκόσμιο επίπεδο. Στη συνέχεια είδαμε ότι τα μέτρα δεν είναι τα ίδια, δεν υπάρχει εναρμόνιση και δεν εφαρμόζονται καν. Ε, και ότι υπάρχουν συμφωνίες γενικές στις περισσότερες περιπτώσεις ε, με ανοιχτά πολλά προβλήματα ε, και βλέπετε ότι υπάρχουν πάρα πολλά αποθέματα και πάρα πολλά οικοσυστήματα τα οποία δεν τα διέπει κανένας κανονισμός και δεν τα έχει αναλάβει κανένας οργανισμός. Κοιτάξαμε λοιπόν άλλα διεθνή φόρα όπου μπορούν να αναλυφθούν δραστηριότητες για να καταπολεμηθεί η παράνομη ε, λαθρέα αναρχιαλία. Σήμερα ε, το FAO, το σχέδιο του FAO είναι ε, νομίζω η πρώτη δομή η οποία ε, έχει αναλάβει ένα σχέδιο καταπολέμησης πρόβλεψης ε, και κατάργησης, ε, πάταξης της άναρχης αλίας το 2001. Δυστυχώς όμως ε, αυτό το σχήμα είναι ακόμα σε ένα πλαίσιο ανάληψης ευθυνών, συνειδητοποίησης, δεν έχουμε περάσει στα έργα, είμαστε ακόμα στους λόγους. Για την καταπολέμηση αυτή ξεκίνησε ένα σχέδιο το 1993 για την συμμόρφωση με τις αρχές του FAO, το οποίο διάρκεσε ως το 2003. Και τελικά ε, είδαμε ότι όλα τα κράτη-μέλη που έχουν σημαίες θα πρέπει να λάβουν ορισμένα μέτρα τα οποία θα είναι μέτρα πιστοποίησης της παροχής ε, σημαίων. Ε, ε, θα πρέπει να υπάρχει η ίδια ευθύνη σε αυτόν τον τομέα τελικά η συμφωνία αυτή κατέληξε μια απλή συμφωνία όπου υποσχόντουσαν τα κράτη-μέλη ότι θα αναλάβουν τις ευθύνες τους. Ήταν απλή υπόσχεση. Τον Μάρτιο 2011 μόνο 39 κράτη στον κόσμο ολόκληρο επικύρωσαν αυτή τη συμφωνία του FAO. Δύο χρόνια πριν ε, ο ΕΦΕΟ προσπάθησε να καταρτήσει ένα κατάλογο με διαφορετικό τρόπο αναπτύσσοντας κριτήρια για την υποστήριξη της παροχής σημαίας και προσπάθησε να αναλάβει δραστηριότητες για παράνομα σκάφη τα οποία δεν έχουν, ε, τα, έχουν σημαίες ευκαιρίας. Και η το κάθε κράτος μπορεί να υποστηριχθεί όχι μόνο από την κρατική δομή αλλά και από ανεξάρτητους οργανισμούς. Αυτή ήταν η αρχική ιδέα και εκεί μπορεί να παρέμβει ε, ο ΕΦΕΟ αλλά βεβαίως ε, δεν έχει περατωθεί καν η συζήτηση από αυτό. Ύστερα υπήρξε μια άλλη οπτική γωνία για την καταπολέμηση της παράνομης άναρχης ε, μια συνολική καταγραφή όλων των σκαφών παγκοσμίως, αυτό να γίνει υποχρεωτικά και ε, στην τελευταία συνάντηση, στο τελευταίο σχέδιο του ΕΦΕΟ, στην ημερήσια διάταξη είχε εισαχθεί αυτό το θέμα και τα κράτη αποφάσισαν ε, να καταγράψουν όλα τα σκάφη που ήταν μεγαλύτερα από 24 μέτρα και σε θελούσια βάση για να γίνει να έχει αυτό δεσμευτικό χαρακτήρα αναρωτιόμαστε πώς θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε σε ποιο μέγεθος δεν έχουμε ακόμα συμφωνήσει. Για να καταπολεμηθεί αυτή η παράνομη αναρχελία χρειάζονται και κρατικές συμφωνίες με την, ε, μέσα στα πλαίσια του σχεδίου βεβαίως του, του διεθνούς δικαίου του ΕΦΕΟ. τελικά έχουμε την ανάγκη της εναρμόνισης των πρακτικών και μέχρι σήμερα, όπως σας είπα, μόνο 23 κράτη έχουν επικυρώσει. Έτσι δούλεψε πάρα πολύ σκληρά για πολλά χρόνια ο ΕΦΕΟ πάνω σε αυτά τα προβλήματα και υπάρχει έλλειψη πολιτικής βούλησης των ε, κρατών για την εφαρμογή αυτών των ε, ωραίων ιδεών και των πολύ ωραίων συμφωνιών. Υπάρχει έλλειψη τεχνικών μέτρων και δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστούν οι δραστηριότητες ε, χωρίς αυτά τα τεχνικά μέτρα. Και επίσης πρέπει να, είναι, να, δούμε την δυσκολία πιστοποίησης που υπάρχει για τα σκάφη και υπάρχουν ε, τα περισσότερα κράτη δεν θέλουν ε, πολύ μεγάλη ε, οργάνωση, ρύθμιση ε, σε σχέση με, που να συνάδει με το διεθνές δίκαιο. Τι άλλες λοιπόν δυνατότητες υπάρχουν, τι άλλα βήματα, τι άλλες αρένες, πώς μπορούμε να δράσουμε για να υπάρξει ένας πιο αποτελεσματικός έλεγχος. Ε, υπάρχει βεβαίως ε, το θέμα του ελέγχου του χρηματοοικονομικού μηχανισμού της Γενικής Διεύθυνσης ΜΑΡΕ, η οποία παρέχει προγράμματα, παραδείγματος χάρη στον Ινδικό ωκεανό, στον Δυτικό, Νότιο-Δυτικό Ινδικό ωκεανό, στην Δυτική Αφρική και στο Νότιο Ειρηνικό υπάρχει ένα άλλο πρόγραμμα το οποίο ε, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι μια πολύ θετική πρωτοβουλία την οποία υποστηρίζουμε και η οποία θα αναπτυχθεί. Αλλά πέρα από όλα αυτά είναι σαφές ότι δεν υπάρχουν τα κατάλληλα εργαλεία, διεθνή εργαλεία για να, να αντιμετωπιστεί ένα πρόβλημα που είναι και διεθνές και βεβαίως οικολογικό. Ε, υπάρχουν διεθνείς συμφωνίες αλλά έχουν λίγους υπογράφοντες και λίγους, ε, πολύ λίγοι είναι αυτοί όπως είπαμε που τις έχουν επικυρώσει. Γι' αυτό ίσως χρειάζεται μια εντελώ διαφορετική προσέγγιση. η Νορβηγία παρακίνησε μια σειρά άλλων κρατών σε μία δράση όπου χρειάζονται κανόνες για την αλληλεία, ότι το να μην υπάρχουν κανόνες είναι έγκλημα και ότι πολλές φορές είναι και οργανωμένο έγκλημα γιατί οι μεγάλη δεν απλώς καταχρώνται τις ευκαιρίες να υπεραλλιεύσουν ελάχιστα σε μία ζώνη αλλά πολύ συγκεκριμένα πηγαίνουν με, σημαίες, με πλοία που έχουν σημαίες ευκαιρίες και ε, εγκληματούν. Ε, υπάρχουν τεράστιες εταιρείες πολλών μετόπων που, έχουν σημαίες, που δίδουν σημαίες ευκαιρία και το να, ταυτιστεί, να ταυτιστούν όλα αυτά τα σκάφη είναι κάτι που διαφεύγει πολλές φορές από τις εθνικές αρχές. Γίνεται ένας έλεγχος τους πρέπει να υπάρξει ένας καλύτερο οργανωμένος τρόπος για να ε, ελεγχθούν. Είναι όμως τόσο μεγάλο το κέρδος τους από τα αλλιεύματα που δεν θέλουν να αποσύρουν αυτά τα σκάφη. Ε, επίσης ε, περιγράφεται η περιοχή η αλλιευτική της ΕΕ σαν μια ζώνη η οποία δεν έχει πολύ ψηλό κίνδυνο και έχει μεγάλο κέρδος. Γίνεται λοιπόν παραβίαση των κανόνων εργασίας, διαφθορά, ε, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, ε, πρόβλημα με τα τελωνία και ήδη ο ΙΕ αναγνώρισε ότι υπάρχουν ε, ορισμένες μορφές ε, αυτών των δραστηριοτήτων που μπορούν κάλλιστα να αναγνωριστούν ως οργανωμένο έγκλημα και χρειάζεται να δουλέψουμε στα πλαίσια του σχεδίου του FAO για να ε, γίνουν αυτές οι προτάσεις, για να αναγνωριστεί ως οργανωμένο έγκλημα αυτή η παράνομη ε, λαθρέα αλληλεία. 59 ε, κράτη έχουν πάρει μέρος σε αυτή την σύμβαση που την έχουμε και ε, που έχει εγκριθεί και χρειάζεται να αναλάβει δραστηριότητες μιας ε, εφιούς έρευνας σε διεθνές επίπεδο για να ε, μπορέσουν να, να εξευρεθούν, να ταυτιστούν αυτές οι παράνομες λαθρές άναρχες δράσεις. Υπάρχει επίσης η Europol, η Interpol που μπορεί να συνεργαστεί. Ένα εμπόδιο είναι ότι πολλές χώρες δεν θεωρούν ότι είναι εγκληματική ενέργεια της παράνομης αλίας, αλλά ότι είναι ένα παράπτωμα μόνο. Ε, η παραβίαση όμως των κανόνων αλίας δεν είναι έγκλημα, αλλά όλο το θέμα της απάτης είναι ε, παράνομο έγκλημα, γιατί μπορεί να χρησιμοποιηθεί βάση του διεθνούς δικαίου ε, αυτό το στοιχείο και θα μπορούσε να συμπεριληφθεί έτσι η συνεργασία της Interpol. Υπάρχουν και άλλες ορισμένες ιδέες σε αυτό το κείμενο του τι μπορεί να πράξει η Ευρωπαϊκή Ένωση και πραγματικά είμαι πολύ περίεργη να ακούσω και τις δικές σας απόψεις ε, και των σκιωδών εισηγητών αργότερα που θα λάβουν το λόγο. Μία φορά πάντως ε, εξετάσαμε την ανάγκη μιας ανεξάρτητης αξιολόγησης ε, για, τα, για την απόδοση των SMOs ε, για να μπορέσουμε να αναλάβουμε δραστηριότητες ε, που αυτό θα αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό βήμα. Τώρα πώς θα μπορέσουμε να πιστοποιήσουμε κάτι τέτοιο. Υπάρχουν οργανώσεις που έχουν στόχο την διατήρηση των αλλιευμάτων, των αποθεμάτων της αλίας. Ναι, αλλά ποιος αλλιεύει. Ε, και φτάσαμε σε μια χρονική στιγμή όπου ε, γίνεται πλέον κατανοητό ότι ε, η κατάσταση των ωκεανών είναι πάρα πολύ σημαντική για την ευμάρεια του πλανήτη ολόκληρου και για τη δυνατότητα ενός μέλλοντος που έχει κάποια ε, τροφική ασφάλεια, δηλαδή για τις επόμενες γενναίες. Ε, και χρειάζεται μεγαλύτερη συνειδητοποίηση. Μιλήσαμε ήδη για την συνειδητοποίηση της κληρονομιάς που αποτελούν οι ε, ωκεανοί για την ανθρωπότητα. Δεν είναι μόνο ένα τυχαίο εμπορικό αποτέλεσμα ή κέρδος το ε, οποίο όταν βλέπουμε πόσο γρήγορα μειώνονται τα αλλιευτικά αποθέματα και πώς καταστρέφεται το οικοσύστημα και ποιες είναι οι δυνατότητες των μελλοντικών γενεών να έχουν τρόφιμα, τρόφιμα πάνω στο τραπέζι τους. Έτσι λοιπόν χρειάζεται μία αξιολόγηση ανεξάρτητη των αλλιευμάτων και νομίζω ότι ο ΙΕ μπορεί να αναλάβει αυτή τη δράση και ε, πιστεύουμε ότι δεν μπορούμε πλέον να περιμένουμε για τον, ε, να περιμένουμε τον FAO να δράσει. Δεν είναι δυνατόν. Χρειάζονται διμερείς δραστηριότητες, χρειάζονται συμφωνίες με μεγάλες αλληλευτικές χώρες, με μεγάλες αγορές καταναλωτών που έχουν μεγάλη επίπτωση στα είδη των ψαριών τα οποία επιτρέπεται να εισαχθούν στην αγορά. Δηλαδή πρόκειται βασικά για τις Ηνωμένε Πολιτείες και την Ιαπωνία. Χρειάζεται ένας συνασπισμός των όσων επιθυμούν να συνασπιστούν ούτως ώστε να ε, υπάρξουν κανόνες για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές και για όλες τις δραστηριότητες, τις αλληλευτικές. Εάν είναι αλήθεια ότι το 20% ε, της ε, παγκόσμιας αγοράς είναι με παράνομη αλληλεία και λαθρέα, πρέπει να να δράσουμε γιατί αν ξέραμε ότι 20% ήταν ελεφαντοστού ή ε, πετρέλαιο ή τι θα κάναμε, τι θα έκανε η ΠΟΕ. Ε, θα πρέπει δηλαδή να υπάρχουν δυνατότητες αυτό το πρόβλημα να το θέσουμε και μέσα στα πλαίσια του ΠΟΕ για να δούμε ε, αν, αν όντω καταλαμβάνει το 20% η λαθρεαλία. Και υπάρχουν τελικά και μερικές τεχνικές ιδέες και δυνατότητες για την επέκταση την επέκταση των ε, διαφόρων ελευτικών τομέων, διάφορες απόψεις που άκουσα ε, στην Ίσπρα ε, θα χρειάζεται να καταρτιστεί μου είπαν μία βάση για την DNA των ηχθείων όχι των αλλιέων των ηχθείων και από πού προέρχονται αυτά τα ψάρια και θα ήταν μια πολύ καλή βάση για να μπορεί να γίνει έλεγχος για την εγκληματικότητα, ε, της παραβιάσης, τι απάτης και κτλ. Ε, παρακαλώ τώρα θα ήθελα να ακούσω τα σχόλιά σας, τις προτάσεις σας. Ε, πιστεύω ότι για την ώρα φαίνεται αδύνατο να καταπολεμήσει κανείς την λαθρεαλία που είναι ένα διεθνές τεράστιο πρόβλημα. Αλλά νομίζω ότι το μόνο, ε, έχουμε όλα τα τεχνικά μέσα, αλλά λείπει η πολιτική βούληση, είναι το μόνο που απουσιάζει. Ε, ευχαριστώ πολύ κυρία Λόβεν για αυτήν την τεράστια εργασία που επιτελέσατε. Πραγματικά. Θα ευχαριστήσω. είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα τα οποία αντιμετωπίζει η παγκόσμια Ελία σήμερα. Η κυρία Άντρες Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Λόβιν για την εξαιρετική προσπάθεια που κατέβαλε. Πρόκειται για σημαντικό θέμα και πραγματικά δύσκολο. Όπως είπε, το 20% της αλίας, από όσων φαίνεται, φαίνεται ότι είναι παράνομη. Αναφέρονται εδώ τα διάφορα προβλήματα που υπάρχουν που είναι δύσκολο να τα χειριστεί όλα η Επιτροπή Αλίας. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να ζητήσουμε και από το Συμβούλιο και από την Επιτροπή και από τα κράτη-μέλη να συμμετάσχουν σε αυτή την προσπάθεια με πρωτοβουλίες διαφορετικές, διότι ο κατάλογος των λιευτικών σκαφών λέγεται είναι περισσότερα από, πιο μεγάλα από 24 μέτρα και η, καταγραφή τους είναι εθελοντική. Η ανταλλαγή απόψεων, αν είναι δυνατόν, θα μας βοηθήσει. Ξέρω ότι σε πολλές χώρες έγιναν, έγινε καταγραφή και οι κατάλογοι των σκαφών στα Μητρώα είναι δημόσιοι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο επίσης και την Επιτροπή Μεταφορών αφορά. Το θέμα της σημαίας επίσης είναι θέμα αξιολόγησης κάποιας χώρας. Θα ήθελα ε, αναφέρεται εδώ ένας εξωτερικός οργανισμός. Ποιος είναι αυτός που θα κάνει κατά κράτο την αξιολόγηση και κυρίως ποια είναι τα κριτήρια για να μπορέσουν να υπάρχουν ομοιόμορφοι κανόνες για όλες τις χώρες όπως και είναι ο λευτικός Τώρα, το κράτος λιμένας. Εδώ υπάρχει το πρόβλημα των ε, λιμένων όπου έχουμε ελεύθερες ζώνες και δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτήν την περίπτωση. Ένα άλλο θέμα που πρέπει να μελετήσουμε και πάλι είναι πολύπλοκο η καθημερινή, είναι το θέμα των ενεργειών που πρέπει να γίνουν σε κάθε χώρα και σε κάθε λιμένα. Επίσης, ένα άλλο θέμα που πρέπει να αναφέρω και μετά θα δούμε ποιες είναι οι λύσεις που προβλέπετε. Όταν εσείς αναφέρεστε στη λαθρέα και παράνομη αλληλεία, αναφέρεται το λιμάνι των Καραρίων Πάλμας. Ξέρω ότι υπάρχουν ε, κάποιες προφορίες για μια μη κυβερνητική οργάνωση που έκανε μια μελέτη, αλλά υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, όχι μόνο στο Παλμας, αλλά και σε άλλες λιμένες, που είναι η εκφόρτωση ε, κλειστών κοντέινερ, στα οποία ε, περιέχονται ε, ψάρια, αλλά δεν ανοίγονται. Αυτό λοιπόν είναι το πρόβλημα. Αν δεν μπορέσει λοιπόν ε, να ανοίξει ε, το κοντέινερ, είναι σε τράνζιτ. Δεν μπαίνουν αυτά τα αλλιεύματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν να βρεθούν λύσεις για αυτό το πρόβλημα. Ίσως θα πρέπει να ζητήσουμε και τη συνδρομή άλλων επιτροπών. Θα πρέπει όμως να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποτέ δεν κατηγόρησε την Ισπανία, ποτέ δεν υπάρχει καταγγελία ότι η Ισπανία έκανε τέτοιες παράνομες δραστηριότητες ε, εκφόρτωσης παράνομων αλληλευμάτων. Επίσης, εκτός από τις χώρες τις τέσσερις που επικύρωσαν τη συμφωνία, έχουμε την ε, δέσμευση των 27 ε, κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επίπεδο ΦΑΟ. Πρόκειται για μία ψήφο σε επίπεδο ΦΑΟ. Επίσης, εκτός από την ε, καταγγελία που νομίζω ότι δεν είναι λογική, διότι έτσι δακτυλοδεικτούμε κατά μια χώρας, Χωρί να αναφέρουμε σε άλλες χώρες τι γίνεται. Το λιμάνι του Ρότερνταμ, όπου εκφορτώνονται υπό τι ίδιε συνθήκε πολύ περισσότερα εμπορετοποιηματοκιβώτια από αυτά τα οποία φτάνουν στο λιμάνι των Λασπάλμας. Νομίζω λοιπόν ότι γίνεται κάτι το αρνητικό με το να καταδεικνύεται έτσι μια χώρα όσον αφορά τις λύσεις. Με τροπολογίες που θα καταθέσουμε θα βελτιωθούμε τα πράγματα. Εσείς λίγα αναφέρετε για τα θέματα της εμπορικής τυχής. Είπατε τι θα γίνει εάν το 20% της ξυλίας ή το άλλο, άλλο παραδείγμα που ενδιαφέρεται. Φαντάζομαι ότι θα πρέπει τα θέματα τα οποία προανέφερα να τα μελετήσουμε περαιτέρω με την συνδρομή άλλων επιτροπών, από τις επιτροπές Μεταφορών. Απ' την άλλη όμως πιστεύω ότι είναι αναγκαίο να μπορέσει να υπάρξει στην αγορά έλεγχος. Νομίζω ότι το τμήμα που αφορά ε, τις διάφορες εμπορικές δραστηριότητες, το εμπόριο είναι πάρα πολύ λακωνικό και με την ε, συνδρομή σας θα ήθελα να το αξίζουν περαιτέρω. Τώρα, ε, εσείς και αναφέρατε κάτι για το DNA, έγινε λάθος τη μετάφραση. Τι ακριβώς συνέβη. Το DNA είναι κάτι που χρησιμοποιείται, η ανάλυση DNA, για να ταυτοποιήσουμε ένα άτομο όχι ένα είδος αλλιεύματος. Τι γίνεται λοιπόν, εκεί το DNA για δύο ψάρια είναι εντελώ διαφορετικό. Τι, τι ακριβώς θέλετε να πείτε με το DNA. Επίσης, θα συνεργαστώ μαζί σας και για τα προβλήματα που θα μπορούσαν ενδεχομένω να προκύψουν. Για να ε, λυθούν τα προβλήματα που αναφέρεται με την Ισπανία, που φαίνεται σε ενδιαφέρει πάρα πολύ. Η Ισπανία, σύμφωνα με αυτά που λέγονται εδώ για παράνομη αλληλεία, αναφέρεται ότι σε θέματα εκφορτώσεων έχουμε ποσοστό 34%, 60% έχει το Ηνωμένο Βασίλειο, περίπου το ίδιο και η Δανία, είναι και η Δανία όσον αφορά τη χωρητικότητα, το Ηνωμένο Βασίλειο και Δανία. Υπάρχει όμως μια διαφορά. Στην Ισπανία δημιουργούνται πολύ περισσότερες θέσεις εργασίες ε, εκφορτώνοντας λιγότερες ποσότητες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό μας ενδιαφέρει και μας ενδιαφέρει να μην συνεχίσουν οι δραστηριότητες παράνομης αλληλείας και θέλουμε να συνεργαστούμε ώστε να υπάρξει εξυγίανση του τομέα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία. Αντρές Περέα. Ο κύριος Κρίς Ευχαριστώ πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Και εγώ συμφωνώ με τις παρατηρήσεις που κάνατε για την ε, ε έκθεση κυρίας Λέβιν. Η δουλειά των σχεδόν εισηγητών γίνεται πολύ εύκολη. Τώρα, για να επανέλθω στις προηγούμενες παρατηρήσεις. Πριν ε, να κάνουμε κριτική στους άλλους, θα πρέπει να είμαστε ε, εμεί σίγουροι ότι έχουμε νοκοκυρέψει το δικό μας το σπίτι. Θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα καμία ε, κυβέρνηση δεν επωφελείται από τις δραστηριότητες παράνομες αλλίες διότι χάνει χρήματα. Θα πρέπει όμως να αναγνωρίσουμε ότι όλες ε, οι κυβερνήσεις μας είναι νόμιμες, αλλά υπάρχει και το κίνητρο του χρήματος. Πολλές φορές λοιπόν κυκλοφορεί υπόπτος το χρήμα και έτσι υποσκάπτονται κάποιες ε, δραστηριότητες νόμιμες θα μπορούσαμε όμως να σταματήσουμε την παράνομη και την άνορχη αλία. Αν χρειάζεται μπορούμε να επιθεωρήσουμε και να ελέγξουμε σήμερα οποιοδήποτε αλλιευτικό σκάφος. Είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα την αλία παρά για την ξυλία. Αυτό όμως που δεν υπάρχει είναι η απαραίτητη πολιτική βούληση να γίνουν οι αλλαγές που χρειάζεται. Το είπε η κυρία Λέβιν. Το θέμα λοιπόν είναι πώς μπορούμε εμείς να προχωρήσουμε, με ποιες προτεραιότητες Πώς μπορούμε να ηγηθούμε όλων αυτών των προσπαθειών. Τώρα, το σημείο κίνησης θα πρέπει να είναι να μπορέσουμε να συνεργαστούμε με άλλες χώρες που θέλουν να καταπολεμήσουν αυτό το φαινόμενο. Ώστε ή να κάνουμε μία ένωση βελτίστων πρακτικών μεταξύ μας ή να περάσουμε στο επόμενο στάδιο που είναι να προχωρήσουμε τις προσπάθειές μας μέσω των ε, διεθνών βημάτων που υπάρχουν. Τώρα, είναι θέμα βούλησης, το επαναλαμβάνω. Το θέμα είναι ποιος θα αναλάβει την πρωτοβουλία. Θα μπορούσα να πω, θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κομισιό, η Προεδρία, οι κυβερνήσεις. Εγώ θα ήθελα να είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι θα προχωρήσουμε, αλλά ποιον εγκαλούμε για να λάβει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης τις σχετικέ πρωτοβουλίε και να πει: Ακούστε, α νοικοκυρέψουμε τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα χρειαστούμε κανένα δύο-τρία χρόνια τουλάχιστον. Αλλά θα θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι αυτέ οι βέλτιστες πρακτικές ακολουθούνται από τους πάντες. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Κρίστινσεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την κυρία Λέβιν για την εξαιρετική της έκθεση. Πιστεύω πως ε, το έγγραφο αποτελεί μια πολύ καλή βάση για την συζήτηση. Μας λέει ποια είναι τα, ποιες είναι οι ελλείψεις. Ε, συμφωνώ με τον κύριο Ντέιβις. Ε, υπάρχει έλλειψη πολιτικής βούλησης. και η κατάσταση την οποία βρισκόμαστε και αντιμετωπίζουμε. Είναι μια κατάσταση όπου πολλοί δεν θέλουν να εφαρμόσουν τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαχείριση της αλίας είναι ένα ζήτημα πολύ σημαντικό για την καταπολέμηση της πλά. Είναι κάτι το οποίο απειλεί την, τα οικοσυστήματα και την ποικιλότητα. Χρειάζεται να λάβουμε υπόψη ότι και οι αλείς οι οποίοι δραστηριοποιούνται με τρόπο νόμιμο αναγκάζονται να αντιμετωπίσουν μια παράνομη αλληλεία, άρα έναν αθέμητο ανταγωνισμό. Μιλήσαμε επίσης και για παράπλευρα σε επιπτώσεις όπως ε, η διαφυγή πόρων κρατικών ε, από την φοροδιαφυγή όπως ε, και ε, όπως η συγκίτρια μίλησε και για τα προγράμματα διαχείρισης για το, του 2012 αλλά από ό,τι φαίνεται τα προγράμματα αυτά δεν απέφεραν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Η στο πλαίσιο των διεθνών επαφών και σχέσεων χρειάζεται να προωθήσει την επιτήρηση όλων αυτών των αλληλευτικών δραστηριοτήτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να παίξει έναν ενεργό και προορατικό ρόλο ε, ενδεχόμενα προσφεύγοντα και στα αρμόδια δικαστήρια προκειμένου να τηρηθούν οι κανόνες ε, και εφαρμόζοντας ε, και επιβάλλοντας σκληρές κυρώσεις για όσους παραβιάζουν τους κανόνες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σάντσος Πρεσέδο έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τα διαδοχικά έγγραφα που μας παρουσίασε και την έκθεσή της. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό διότι αν υπάρχει κάποια δραστηριότητα που ασκείται παγκοσμίω είναι η αλία. Και είναι δύσκολο να μπορέσει κανείς να χωρίσει την εσωτερική και την εξωτερική πολιτική αλίας. Βασικά διότι η αλία είναι μέλος του κλάδου ειδών διατροφής και τα περισσότερα προϊόντα τα οποία καταναλώνουμε σε τον κλάδο αυτό είναι εισαγόμενα προϊόντα. Διερωτώμε λοιπόν αν και οι υπόλοιποι αλλιεύουν όπως εμείς αλλιεύουμε και θα θέλαμε να ανηλεύουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, πρόκειται για ένα θέμα επιβίωση τη ίδια δραστηριότητα τη Ελία. Θα πρέπει λοιπόν να του προσδώσουμε την μέγιστη δυνατή σημασία. Και θα πρέπει να μπορέσουμε να διαρθρώσουμε την πολιτική μας με τρόπον ώστε και να υποστηρίζουμε την υπεύθυνη και νόμιμη ελία και να μπορούμε με οργανωμένο τρόπο να καταπολεμήσουμε τις παράνομες δραστηριότητες στον τομέα. Γι' αυτό οποιαδήποτε πρόοδος γίνει υπέρ της διαφάνειας και της ε, ανιχνευσιμότητας, ώστε να μπορέσει η διαχείριση του όλου τομέα να γίνεται και βάση επιστημονικών ερευνών και ε, οριζόντια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τις μεθόδους και τα μέτρα που να θα πρέπει να το κάνουμε έχοντας κατά νου ότι θα πρέπει και να βελτιώσουμε τη δική μας αλληλευτική πολιτική και να δώσουμε σημασία στην παγκόσμια διάσταση της δραστηριότητα αυτής. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να συνοδεύσουμε και να υποστηρίξουμε την ΦΑΟ και όλες τις οργανώσεις οικογένειας των Ηνωμένων Εθνών και την δική μας εμπορική πολιτική για να ενεργήσουμε σωστά. Και στην εμπορική πολιτική σε πολυμερές επίπεδο, αλλά όπως πολύ ε, εύστοχα είπαν οι συνάδελφοι και την εμπορική ε, πολιτική την οποία κάνουμε εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχουμε βεβαίως κατά νου την ασφάλεια των ειδών διατροφής που θα μπορούσε να έχει και επιπτώσεις και στην υγεία. Ανιχνευσιμότητα, είπαμε, και έλεγχος. Σε όλα τα πλαίσια της ε, αλλιευτικής ε, αλύση, Πιστεύω λοιπόν ότι Αυτά τα θέματα θα πρέπει να τα προσέξουμε κυρίως και με τις αλληλευτικές ε, συμφωνίες που έχουμε με τρίτες χώρες και ε, γενικότερα με την πολιτική ανάπτυξης. Βεβαίως πρέπει να πω ότι υπάρχει η διάσταση των εξωτερικών σχέσεων ε, που είναι ενδιαφέρουσα. Γι' αυτό λέγω ότι η εργασία που επιτέλεσε η συγγήτρια είναι εξαιρετική. Θα πρέπει να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση και όπως σας είπα δεν μπορούμε να καταπολεμήσουμε την παράνομη αλληλεία αν την αποσυνδέσουμε με την επιβίωση και το μέλλον της νόμιμης αλληλείας. Σας ευχαριστώ. Όπως ανέφερε και η κυρία Λόβιν στις εισαγωγικές παρατηρήσεις, η Νορβηγή... είπαν ότι θα πρέπει να θεωρείται έγκλημα η παράνομη και ελαθρέα αλία. Το πρόβλημα είναι ότι κάποιοι δεν αναφέρονται καν σαν να έχει να, να κάνουμε με μια εγκληματική δραστηριότητα. Περί αυτού όμω πρόκειται. Το ξέρουμε από τις αποδείξεις που υπάρχουν και αυτό επιβεβαιώνεται και στον έγγραφο της κυρίας Λόβιν. Όντως, πρόκειται για οργανωμένο έγκλημα που επιτελούν γκάγκστερ παγκοσμίων. Και ξέρουμε ότι εδώ διακινούνται τρομερά ποσά. Και πολύ και ξέρουμε επίσης ότι υπάρχει καταστροφή του περιβάλλοντος, κατάχρηση των ε, εργαζομένων, ε, χρησιμοποίηση επικινδύνων αλλιευτικών σκαφών και έχουμε εδώ αποδείξεις αλλιευτικού σκάφους των οποίο υπήρχαν πάνω 200 ε, ε, εργαζόμενοι που δούλευαν στιβαγμένοι σαν σαρδέλες και σε πακέτο με συνθήκες τρομερές. Και όλα αυτά για να μπορέσουν να εργαστούν με στη νύχτα παράνομα και μυστικά και πολλές φορές με, την, με συνεργούς άλλων αλλιευτικών σκαφών για να μπορέσουν να διοικητεύσουν τα αποτελέσματα της παράνομης δραστηριότητάς Υπάρχουν ε, λοιπόν τρομερά εγκλήματα που γίνεται εις βάρος όλων των των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε όντως με διαφθορά, με απάτη σε διεθνές επίπεδα και θα πρέπει όντως να αναλάβουμε ηγετικό ρόλο για την καταπολέμηση αυτού του προβλήματος και όντως θα πρέπει να αναγνωριστεί αυτή η δραστηριότητα ως εγκληματική και να επιμείνουμε ώστε να δημιουργηθεί πρώτα απ' όλα ένα παγκόσμιο μητρό στο οποίο θα καταγράφονται αυτά τα παράνομα αλλιευτικά σκάφη. Και μπορούμε να κατανοήσουμε ότι υπάρχει αντίδραση και αντίσταση και το να προχωρήσουμε καταρχάς με ένα εθελούσιο σύστημα καταγραφής τους ε, είναι εντελώς άχρηστο. Είναι άχρηστο κυρίως για τα αλλιευτικά σκάφη που έχουν ε, μήκος περισσότερο από 20-24 μέτρα. Ξέρουμε ότι υπάρχουν χώρες που προσπαθούν να αποκρύψουν τα σκάφη και τις δραστηριότητε αυτές και θα πρέπει να τις ονοματίσουμε, να τις ξέρουν όλοι. Διαφορετικά θα συνεχίσουμε με αυτή την ε, ε, καταχρηστική δραστηριότητα μέχρι που θα καταρρεύσει η αλληλευτική δραστηριότητα για κάποιες χώρες. Παρακαλώ η κυρία Γιόλσεν από την Κομισιόν, τη Γενική Διεύθυνση ΜΑΡΕ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι θα ήθελα και εγώ απλώ και μόνο να επαναλάβω ότι είναι πολύ καλή αυτή η έκθεση. Περιμένουμε την οριστική, αλλά πρέπει να πω ότι μας ικανοποιεί απόλυτα αυτή η έκθεση. Όπως... Ξέρετε, δεν έχουμε φτάσει στο τέλος του αγώνα μας, πρόκειται όμως για ένα περαιτέρω βήμα, για μια περαιτέρω βοήθεια για να μπορέσουμε κάτι να κάνουμε για την πρόσφυση της νόμιμης αλλίας. Όσον αφορά το οργανωμένο, σύμφωνα με την κυρία Λέβη, είναι πάρα πολύ σημαντικό να θεωρηθεί όντως ως έγκλημα. Πρόκειται για εγκληματική ενέργεια και κλοπή των αλλιευτικών πόρων. Νομίζω ότι ούτως ή άλλως πριν ε, να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι σε διεθνές επίπεδο θα πρέπει να υπάρχει και η βελτίωση της σχετικής εθνικής νομοθεσίας. Και πραγματικά αυτό θα ήταν χρήσιμο αν υπήρχε μια τέτοιου είδου πρόνοια εκ μέρους όλων των κρατών μελών. Με συγχωρείτε, το σημειώσουμε γιατί κυρίως δεν ασχολούμαι εγώ με αυτά τα θέματα. Επίσης έχουμε την δυνατότητα μέσω των νέων κανονισμών να κάνουμε και σε εθνικό επίπεδο κάποιες έρευνες και να ενθαρρύνουμε και άλλους διεθνείς και άλλα διεθνή συμβαλόμενα μέρη να ενεργήσουν τον ίδιο τρόπο. Το πρόβλημα είναι ότι στις διεθνείς αγορές πρέπει να πούμε ότι και εμείς ως κοινότητα έχουμε αλλιευτικά σκάφη με κοινοτικέ σημαίε ευκαιρία. Άρα θα πρέπει και αυτό το θέμα να το εξετάσουμε και να το λύσουμε εμεί πρώτα στο δικό μα επίπεδο. Σα ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε, κυρία Γιόνσεν, η συγγήτρια, κυρία Λέβιν. Ευχαριστώ για τα ενδιαφέροντα σχόλιά σας. Θα προσπαθήσω να απαντήσω με τη σειρά. Κυρία Μπαρέα, με ρωτήσατε ποιες θα είναι οι οργανώσεις που μπορούν να κάνουν την αξιολόγηση για το θέμα των σημεών. Ο ΦΑΟ έδειξε αυτό το ζήτημα πρώτος. Εάν ε, χώρα σημαία ε, κάνει την αξιολόγηση από μόνη τη. Ε, αυτό μπορεί να είναι σημαντικό, αλλά θα πρέπει να έχουμε κριτήρια τα οποία θα ισχύουν ε, παγκοσμίω. Νομίζω ότι το FMO είναι το καταλληλότερο φόρουμ που θα μπορούσε να αναλάβει κάτι τέτοιο. Ίσως όμως θα χρειαστεί η συγκρότηση ενός νέου φόρουμ για την αξιολόγηση και για την εφαρμογή των ε, βέλτιστων προτύπων. Τώρα το ζήτημα των νήσων ε, λασπάλμας. και των Καναρίων Ίσων. Ναι, και άλλα λιμάνια όντως εντοπίστηκαν ε, που έχουν αυτές τις δραστηριότητες ε, στα λιμένες τους. Υπάρχουν διάφορες ε, με κυβερνητικές οργανώσεις που έχουν παραπονεθεί. Τώρα το Δεν ξέρουμε κατά πόσον ε, ο λιμένας της Λαπάλμας έχει βελτιώσει και αυξήσει τους ελέγχους αναφορικά με την παράνομη, με την και λαθρέα αναρχιαλία. Όντως ε, είναι ένα μεγάλο σημαντικό λιμάνι των Λασπάλμας. Ε, εντάξει, άκουσα το σχολείο σας για το Ρότερδαμ και για τα εμπορευματοκιβώτια που βρίσκονται υπό διαμετακόμιση εκεί. Τώρα για τους περαιτέρω ελέγχους στις αγορές συμφωνώ απόλυτα. Ναι, όντως δεν αποδώσαμε ιδιαίτερη προσοχή στο έγγραφο, αναφέραμε μόνο τον ΠΟΕ, αλλά θα λάβω υπόψη μου την πρότασή σας Νομίζω πως υπάρχουν πολλές ομοιότητες με την έκθεση Καντέκ και για τα υψηλά πρότυπα που θα πρέπει να εφαρμόζουμε. Τώρα το κατάλογος σχετικά με τα αλλιεύματα είναι μια καλή ιδέα. Τώρα τα κράτη και το ζήτημα των σημείων. Τώρα για το DNA ίσως να έχετε δίκιο. Εγώ πρότεινα να γίνει ένα γενετικό μητρό έτσι ώστε να μπορούμε να εντοπίζουμε διάφορες ποικιλίε εχθείων και να τις ε, ταυτοποιούμε με κάποιες βιολογικές αναλύσεις αν θέλετε να δούμε λοιπόν κατά πόσον ε, το DNA ναι, ναι, δεν είναι ο κατάλληλος όρος. Μάλλον έχετε δίκιο. Τώρα ο Chris Davis, το να βάλουμε ε, να βάλουμε τα, να φτιάξουμε τα πράγματα στην οίκο μας. Ε, ναι, έχεις ε, δίκιο. Αν θέλουμε να είμαστε όμως αξιόπιστοι διεθνώς, χρειάζεται να βελτιώσουμε τις προσπάθειές μας στο ζήτημα των ελέγχων και να πείσουμε ότι τα κράτη μας πρώτα απ' όλα ε, καταπολεμούν και δεν ε, εφαρμόζουν την πλά. Εγώ είμαι Σουηδή και μπορώ να πω δίχως τύψεις ότι η Κομισιόν θεώρησε πως 23% τον γάβο που αλευόταν στα σουηδικά ύδατα ήταν παράνομος. Τώρα ε, αυτό το ποσοστό έχει μειωθεί κατά 8-9%. Αλλά με υπάρχει. Άλλα κράτη φυσικά τα έχουν πάει χειρότερα, άλλα καλύτερα από μας, ε, αλλά είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να μας αποσχολήσει σε όλα τα ενωσιακά γραμμή. Χρειάζεται να γνωρίσουμε ότι 60% των αλλιευμάτων που καταναλώνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ξέρουμε ότι αλλιεύεται νομίμως of the willing. Το 60% λοιπόν είναι εισαγόμενο. Τώρα η ιδέα του Chris Davis ε, είναι καλή. Αν θέλουμε να προχωρήσουμε τάχιστα, διότι αν δούμε το ιστορικό της ΦΑΟ και άλλων οργανισμών όπως τα FMOs, παρατηρούμε ότι προχωρούν και ενεργοποιούνται με μεγάλη καθυστέρηση. Η Ιαπωνία είναι ένας ε, καλό εταίρος, η Αυστραλία επίσης, αλλά να προχθώσουμε να πάρουμε το μέρος μας και την Κίνα, τότε αυτό θα είναι μεγάλη επιτυχία. Χρειάζεται λοιπόν να προχωρήσουμε και πιστεύω πως η Κομισιόν μπορεί να αναλάβει το ηγετικό ρόλο και να ακολουθήσει το Συμβούλιο Υπουργών. Ευχαριστώ κύριε Σάντερσεν για το σχόλιο σας. Ναι, όντως πρόκειται για αθέμητο ανταγωνισμό όταν επιτρέπουμε σε παράνομα προϊόντα να ανταγωνίζονται νόμιμα προϊόντα. Εμείς προσπαθούμε να ε, ε, δημιουργήσουμε αποθέματα και έρχεται κάποιος και μας κλέβει τα, τα αποθέματα αυτά, τα λιεύματα, ε, εξοντώνει το γόνο κλπ. Χρειάζεται λοιπόν ε, να εξετάσουμε το θέμα των σχέσεών μας ε, με τις αναπτυσσόμενες χώρες. Ε, αυτό απαιτεί μια σφαιρική προσέγγιση και εμπίπτει στο, στο πλαίσιο της ανδρυσιακής πολιτικής, κύριε Πρεσέντο. Ναι, όντως η αλληλεία είναι μια παγκόσμια δραστηριότητα και ίσως ε, να είναι η πρώτη πραγματικά παγκόσμια δραστηριότητα. Δεν γνωρίζει σύνορα, αλλιεύονται σε, ένα, σε μια ζώνη και εισέρχονται και εκφορτώνονται σε άλλες περιοχές, σε άλλα λιμάνια κλπ. Εντάξει, εδώ εμπίπτει και το ζήτημα της ε, ασφάλειας των τροφίμων. Ε, τονίσατε την σημασία του εμπορίου. Κύριε Στίβενσον, σχετικά με την ΦΑΟ, οργανώσατε ένα hearing, μια κρόαση για την καταπολέμηση της παράνομης ε, αλίας και κατά πόσο πρόκειται για οργανωμένο έγκλημα. Ναι, η ΦΑΟ είναι ένα διεθνές όργανο το οποίο εξετάζει το ζήτημα αυτό εδώ και χρόνια. Πάντως σε κανένα από τα έγγραφα της ΦΑΟ δεν αναφέρεται ο όρος έγκλημα. Πρόκειται για μια παρατυπία, για μια παράβαση, παράβαση κανόνων κλπ. Αλλά όχι έγκλημα. Μιλάμε για δέκα δις ευρώ ετησίως που ληστεύονται από τις θάλασσες. Πρόκειται για ένα τεράστιο οικονομικό έγκλημα και είναι και περιβαλλοντικό έγκλημα επίσης αλλά ε, οι περισσότεροι είναι ευαίσθητοι στην οικονομική πτυχή του εγκλήματος. Θα πρέπει να πούμε στην ΑΝΤΟΚ, την Παγκόσμια Οργάνωση πολέμηση Εγκλήματος, να ασχοληθεί με το ζήτημα. Ευχαριστώ και την Κομισιόν για τα ενθαρρυντικά σας λόγια. Ευχαριστώ. Yeah, λοιπόν, για το δεύτερο έγγραφο που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Νομίζω ότι πράγματι προχωράμε και να σου το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε για την καταπολέμηση της ΠΛΑ. Στις 24-25 Μαΐου θα συζητηθεί 12-13 Ιουλίου θα ψηφίσουμε τις τροπολογίες, 19 Σεπτεμβρίου ε, στην, Επιτροπή μας και στην Ολομέρη θα περάσει από την δεύτερη σύνοδο του Οκτωβρίου. Λοιπόν, τον Ιούλιο θα εξετάσουμε τις τροπολογίες. είναι, ποια ήταν η προθεσμία για την των τροπολογιών. Δεν ε, το είπαμε ακόμα, αλλά ανταλλαγή απόψεων επί των τροπολογιών θα είναι 12 και 13 Ιουλίου. Η έκθεση 24-25 Μαΐου ήταν έτοιμη και τότε θα ε, μιλήσουμε για την προθεσμία κατάθεση τροπολογιών. Θα είναι κάπου τέλη Μαΐου, αρχές ε, Ιουνίου. Ε, τέλη, τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου. Και τώρα να περάσουμε στο σημείο 10 της μέσης διατάξεως. Ε, το οποίο αφορά την συνάντηση που είχαμε στη Ρώμη και επρόκειτο να συζητηθεί στην 25 Μαρτίου αλλά ανεβλήθη και έτσι Φυσικά εδώ δεν ε, φταίει η κυρία Λόβιν, ε, η οποία είχε μεταβεί στην Ρώμη, είχε συμπεριληφθεί στην επίσημη ψηφία της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και είχε μεταβεί ως παρατήδρια στην Ρώμη και τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Λόβιν για να μας αναφέρει σχετικά με την συνεδρίαση. Ευχαριστώ πολύ και κυρίως που με ακούτε τόση ώρα να μιλώ και θα συνεχίσετε να με ακούτε. Θα προσπαθήσω να εξηγήσω τι συνέβη στη Σύνοδο Επιτροπής Αλίας Κόφη. Ε, καταρχήν η ε, FAO που είναι η Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών ε, για την ε, On fisheries under the... και τρόφιμα ε, ε, υπό την αιγίδα της ΕΦΑΙΟ λοιπόν ε, έγινε αυτή η συνάντηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έγινε πλήρως, πλήρες μέλος της ΚΟΦΗ το 1993 και τα διάφορα κράτη-μέλη ήταν το καθένα πλήρες μέλος ξεχωριστά προηγουμένως. Πριν από κάθε συνεδρίαση γίνεται μια ανάλυση της ε, ημερήσιας διάταξης, ποια θέματα είναι ε, στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ποια θέματα είναι στην αρμοδιότητα των κρατών μελών για να μπορέσουν να υπάρξουν ψηφοφορίες. Δεν μπορούσαν όλοι να μιλήσουν στην συνεδρίαση όλοι οι εκπρόσωποι της ΕΕ. Οι προτεραιότητες της Επιτροπής Αλίας είναι η προαγωγή της διατροφικής ασφάλειας, οι αηφόροι κανόνες εξέλιξης, η ανάγκη διαχείρισης και η στατιστική συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών. Αυτό είναι ο στόχος καταρχήν της Επιτροπής, ε, ο πολύ σημαντικός ε, Αλίας. Ε, είχα πάρει μέρος ε, ως εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ήταν παρόν ένας εκπρόσωπος ε, των Πρασίνων και η κυρία Μάνια Κράσκο που ανήκε στη Γραμματεία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Μαριλία για την εξαιρετική εργασία, για την συγκέντρωση των στοιχείων, για την έκθεση την οποία βασίζομαι τώρα που είναι πραγματικά χρήσιμη. Με βοήθησε. Ο, ο κύριος Αντώνιο Φερνάρες ήταν ε, από τη Γενική Διεύθυνση ΜΑΡΕ, διεύθυνε την, τις ε, συνομιλίες και έγινε μια συζήτηση για το κατά πόσο μπορεί το Κοινοβούλιο να συμμετέχει σε διεθνείς συνεδριάσεις και φόρα ε, χωρίς να έχει ε, τις αρμοδιότητες που ασκεί βάσει της συνθήκης της Λισαβόνας. Ε, για την... <clears throat> Υπάρχουν ορισμένες, ορισμένοι κανόνες της οργάνωσης κόφη, τους οποίους θα σας διαβάσω. Καταρχήν είπαμε ότι χρειάστηκε μια ανεπίσημη ανταλλαγή απόψεων ε, εμείς ε, ήμασταν παρόντες ως ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά όχι στις επίσημες συνεδριάσεις εκεί όπου ελαμβανόντουσαν οι αποφάσεις. Το, τα θέματα που ήταν προβληματικά για την Ε ήταν τρία. Αν τα κράτη-μέλη πρέπει να καθορίζουν τα μέλη μέχρι την τελευταία στιγμή, καταρχήν το θέμα των, ε, της ε, παράλληλης αλλίας. Technical guidelines and the EU... Το θέμα των απορρίψεων και των παράπλευρων και ε, αρχικά δεν έγινε η έγκριση των κατευθυντήριων γραμμών πάνω σε αυτό το σημείο. Δηλαδή η συζήτηση για την ε, ευρωπαϊκή, για ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το τομέα δεν είναι ακόμα όριμη, δεν είναι ακόμα έτοιμη και γι' αυτό δεν ε, εγκρίθηκαν οι κατευθυντήριες γραμμές σε επίπεδο FAO. Ένα άλλο θέμα που που προκάλεσε αντιθέσεις είναι το θέμα των διεθνών κατευθυντήριων γραμμών για τις ε, μικρής, αλίες, μικρής κλίμακας αλίες. Κάτι το οποίο χρειάζεται τεχνικής φύσεως ε, κατευθυντήριες γραμμές για τα μικρά σκάφη και για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Εκεί δεν υπήρξε συμφωνία των περισσότερων κρατών μελών της ΕΕ. Αν θα υποστήριζαν αυτή τη θέση όχι. Και τελικά υπήρχε ε, και ένα λιγότερο αντιφατικό θέμα, αλλά με πολλή συζήτηση για τη χρηματοδότηση του της ε, ε, οικολογικής αλίας, τι ποσό, τι συνολικό ποσό χρειάζεται να διατεθεί για να μπορέσει να υπάρξει σωστή χρηματοδότηση του σχεδίου. Επίσης, οι μοιρασμένε αρμοδιότητες με την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, μοιράζονται ε, ως εξής μπορεί ως η Ευρωπαϊκή Ένωση ως ε να λάβει το λόγο και όχι τα κράτη-μέλη μεμονωμένα Επίσης υπήρξε το θέμα των αρμοδιοτήτων, της εκλογής των αρχαιρεσιών, έγινε εκλογή Προέδρου και τα υπόλοιπα ε, για την επόμενη, αφέθηκαν για την επόμενη συνεδρίαση. Ε, ήταν 15 κράτη-μέλη ε, παρόντα και υπήρχαν και παρατηρητές δηλαδή 64 διακυβερνητικές οργανώσεις και μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες είχαν λόγο, είχαν τη δυνατότητα να λάβουν το λόγο. Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης ήταν η, ο κώδικας συμπεριφοράς για, για την υπεύθυνη αλία. Ε, ήταν μια πάρα πολύ θετική συμφωνία. Αυτός ο κώδικας συμπεριφοράς ε, θα ήταν πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ θετικός ε, αν υπήρχε εφαρμογή του. Αν υπήρχε σωστή εφαρμογή του δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Ε, όμως όπως δεν εφαρμόζεται, αυτό που συζητήθηκε στο σημείο αυτό της ημερήσιας διάταξης ήταν να υπάρξει ένα ερωτηματολόγιο το οποίο είχε αποσταλεί στα κράτη-μέλη και ρωτούσε ποια ήταν η πρόοδος των εργασιών, η πρόοδος της εφαρμογής αυτού του κώδικα συμπεριφοράς για την υπεύθυνη αλληλεία ε, και τα κράτη απάντησαν, ε, όχι όμως όλα, μόνον 16 και ήταν μικρή η συμμετοχή, πραγματικά είναι απογοητευτικό το να τη διαπιστώνουμε και υπήρξε σχολιασμός από όλες τις χώρες που έπαιρναν μέρος ε, Δηλαδή είναι μικρό το ποσοστό των κρατών που ε, πήραν μέρος στις, στις, απαντήσεις ενώ όλοι έχουν αλία και αυτό σημαίνει ότι δεν παρακολουθούμε την πρόοδο, δεν υπάρχει πρόοδος και άρα δεν εξελισσόμεθα με ταχύτητα. Ε, ε, για τον κώδικα συμπεριφοράς επίσης έχετε το διεθνές σχέδιο δράσης, τις στρατηγικές, έχετε το θέμα των καρχαριών, των υπερβολικών αλλιευμάτων, ένα διεθνές σχέδιο της καταπολέμησης λαθρέας ε, ε αλλά όλα αυτά είπαμε ότι δεν εξελίσσονται πολύ γρήγορα. Αυτά περί του πρώτου σημείου. Δεύτερο σημείο ήταν οι αποφάσεις και της υποεπιτροπής για το, την αλληλεία, για το εμπόριο των ηχθείων ε, και την υδατοκαλλιέργεια. Υπήρξαν γενικές κατευθυντήριες γραμμές και σε αυτόν τον τομέα και δεν υπήρξαν κράτη-μέλη που να πάρουν ατομικά τον λόγο μέσα στα πλαίσια της, ε, του FAO. Μίλησαν για την επίπτωση στο διεθνές εμπόριο, ε, την ανάγκη των κατευθυντηρίων γραμμών και οι αναπτυσσόμενες χώρες που πήραν το λόγο πρέπει να πω ότι πάντα, κάθε φορά, ανησυχούσαν για την ε, οικονομική επίπτωση που θα είχε αν εφαρμοζόντουσαν αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές όντως. Το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη ήταν η πρόοδος που έγινε σε σχετικά με μέτρα κατά της παράνομης ε, ε, και άναρχης αλίας ε, και όλα αυτά ήταν ειδικού ενδιαφέροντος για μένα εφόσον είναι το θέμα με το οποίο ασχολούμαι και ανάφερα ήδη ότι υπάρχουν ε, ορισμένα μέτρα τα οποία αφορούν τους κρατικούς λιμένες, το θέμα ε, των σημεών ευκαιρίας και ε, των επιδόσεων στον τομέα των σημεών, τα, σχέδια, τα μέτρα που έχουν σχέση με τις αγορές. Υπήρξε μεγάλη, μεγάλη υποστήριξη για το θέμα της, του Γενικού Μητρώου και η Ζηλανδία, η Αυστραλία, η ΙΠΑ, μας υποστήριξαν καθώς και η Ιαπωνία σε ό,τι αφορά αυτό το σχέδιο. Μετά πήρε το λόγο η Κίνα και είπε όχι. Πιστεύουμε ότι χρειάζεται μια πιο σταδιακή προσέγγιση σε θελούσια βάση και η Ινδία επίσης στη συνέχεια πήρε το λόγο και συμφώνησε με την Κίνα και έτσι περατώθηκαν οι διαδικασίες. Θα υπάρχει λοιπόν ένα μητρό αλλά σε θελούσια βάση. Αυτό, αυτή είναι η απόφαση που ισχύει για την ώρα. Θα δούμε που θα πάμε στο μέλλον με βάση αυτή την πρώτη απόφαση. Στη συνέχεια υπήρξε το θέμα ε, αλληλεία και υδατοκαλλιέργεια και κλιματική αλλαγή. Η διαχείριση των ηχθείων μαζί με το θέμα της βιοπικιλότητας. Ε, και έγινε μεγάλη συζήτηση και όπως είπα υπήρξαν ορισμένες αντιφάσεις μέσα στην αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην τελευταία στιγμή δεν συμφώνησαν αν θα πρέπει να προσυπογράψουν αυτές τις ε, κατευθυντήριες γραμμές. Οι Ηνωμένε Πολιτείες είπαν ότι θα έπρεπε, ναι. Ε, εμείς δεν αποφασίσαμε ε, το αν ήταν από χρόνο λόγος για να μην τις εγκρίνουμε αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές. Ύστερα μιλήσαμε για, τις, ε, για την αλία μικρής κλίμακας, ένα επόμενο ε, σημείο στην ημερήσια διάταξη και αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές τις ε, υποστήριξε η ΕΕ μετά από συζήτηση μεταξύ των μελών. Και το τελευταίο σημείο ήταν οι προτεραιότητες για το 2012 και το 2013 αυτά που συμφωνήθηκαν ήταν να συνεχίσουμε να δουλεύουμε, να υπάρχει συναγωγή πληροφοριών ε, σε αυτή τη φάση, όσο περισσότερες πληροφορίες μπορούμε και να ε, ασχοληθούμε με τη διαχείριση των τεχνικών προδιαγραφών για την αλία μικρής κλίμακας, για την μείωση ε, των αλλιευμάτων και τα, των, της υπερβολικής αλίευσης κτλ. Ε, τελικά οι μέρες ήταν πολύ φορτωμένε με συνεδριάσεις, με πολλή εργασία, με πολλούς ομιλητές, ε, διάφορες μη κυβερνητικές οργανώσεις, 64 στον αριθμό. Η συνολική εντύπωση ήταν ότι υπήρξε μια πολύ βραδία εξέλιξη γενικότερα στο θέμα και ειδικά οι αναπτυσσόμενες χώρες ζητούν κάθε φορά περισσότερη τεχνική βοήθεια και στήριξη και, δεν, και εφαρμόζουν τις χρηστές αποφάσεις ε, και αυτό είναι φαίνεται το μείζον πρόβλημα. Τελικά λείπει πάλι, απουσιάζει η πολιτική βούληση και εδώ το διαπιστώνουμε γιατί υπάρχει τόσο δισταγμός ορισμένων κρατών όπου δεν θέλουν να προχωρήσουν περισσότερο, να εξελιχθούν σε αυτόν τον τομέα. Αυτά κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, κυρία Λόβεν για την πληρέστατη έκθεσή σας αλλά και για τη βοήθειά σας. Ε, ε κύριε Λόβεν, θα ακούσουμε τώρα τα μέλη. Δεν βλέπω όμως κανένα να σηκώνει το χέρι του. Ίσως να ήταν όλοι πάρα πολύ ευχαριστημένοι από τα στοιχεία που φέρατε και ίσως μπορώ να πω ότι θα ξαναβρεθούμε στις 3 το απόγευμα σε κλειστή συνεδρίαση για μια ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή Αλίας που αφορά τις συμφωνίες με τις τρίτες χώρες και τις σχετικές διαπραγματεύσεις και στη συνέχεια θα ξανανοίξουμε τη συνεδρίαση για να υπάρξει ανταλλαγή απόψεων με τον Ευρωπαίο Συντονιστή ε, ο θα γίνει μια συνεδρίαση συντονιστών νωρίτερα από ό,τι έχει προβλεφθεί, μάλλον αυτό ε, προβλέπουμε και ελπίζω όλοι οι συντονιστές να είναι παρόντες εδώ για την απογευματινή συνεδρίαση ή τουλάχιστον να προσπαθήσουν γύρω στις 4.30. Ε, θα, θα τα πούμε το απόγευμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.